Αφήστε συνάδελφοι, παρακαλώ πάρτε τις θέσεις σας. Euh, λοιπόν, ξεκινάμε, η οποία έχει η συνάντησή μας η σημερινή ένα έκτακτο χαρακτήρα. Ε, βασικά αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα είναι η τροποποίηση του, ε, του νέου πλαισίου, του χρηματοδοτικού πλαισίου και κυρίως ε, τίθεται το θέμα της ε, απλοποίησης και σε ποιο βαθμό μπορεί κάτι τέτοιο να αναζωογονήσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Ξέρετε ότι έχετε μάλλον την ημερήσια διάταξη, δεν έχω παρατηρήσεις πάνω σε αυτό, δεν έχω να κάνω ανακοινώσεις γιατί προηγήθηκε μια συνάντηση των συντονιστών της Επιτροπής Προϋπολογισμών για τις συστάσεις ε, για τον προϋπολογισμό 17. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό αύριο στις 9 το πρωί. Θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε ότι τα πρακτικά, τα τελευταία που έχουν διανεμηθεί τις 23ης και 24ης Μαΐου δεν δημιουργούν πρόβλημα. Οπότε μπορούμε, κυρία Συμπρόεδρε, να ξεκινήσουμε τη σημερινή συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση ε, Θέλω να ευχαριστήσω εδώ την κυρία Γκρέσλε για την παρουσία της εδώ σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιτροπές μας να μπορέσουν να λειτουργήσουν ε, ε, εν πλήρη εμπιστοσύνη και με αρμονία. Ο κανονισμός αυτός, έτσι όπως έχει διατυπωθεί, μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα σε επίπεδο εφαρμογής και μπορεί να προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις οι οποίες θα δυσκολέψουν τις επιδόσεις τις οποίες προβλέπουμε. Ξέρετε ότι η Επίτροπος Γεωργίευα εμένει στο θέμα της επίδοσης σε σχέση με τους στόχους. Και έτσι όπως εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτός θα μπορούσε να βλάψει εν πολλής, για να μην πω να καταστρέψει, ε, τις ελπίδες τις οποίες έχουμε σχετικά με τις επιδόσεις. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να διαβουλευτείτε με τους εμπλεκομένους και να δείτε τις σχέσεις που έχουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πραγματικά οι διαδικασίες που έχουν να ακολουθήσουν είναι τρομακτικά περίπλοκες και γι' αυτό υπάρχουν πλέον εμπειρογνώμονες ενδιάμεση επαΐονται σε ενδιάμεση ανάμεσα στους πολίτες, τους επιχειρηματίες και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε η Ευρώπη δεν ομιλεί άμεσα με τους πολίτες της και αυτό δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Κατά συνέπεια λοιπόν η ενδιάμεση αναθεώρηση είναι κάτι το οποίο είναι σαφές ότι θα πρέπει να πετύχουμε με επικοδομητικό τρόπο και ασκώντας κριτική για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά. Η απλοποίηση, η απλούστευση, μας το επενθύμησε η κυρία Γεωργίευα, είναι βασικός της στόχος και γι' αυτό πρέπει να συνδράμουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε περαιτέρω μορφές ε, απλοποίησης. Λοιπόν, ε, μιας και είμαι συμπρόεδρος εδώ, ε, πρέπει να δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αρτή και καλώς ορίσατε όλοι σας. Θα ήθελα στο παρόν workshop ε, να πω ότι συμμετέχω και ω εισηγήτρια για τα θέματα αυτά εδώ και καιρό και θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν ε, το τι έχουμε κάνει και ως τώρα. Και στο θέμα λοιπόν αυτό είμαι σε θέση να μιλήσω για αυτά που έχει κάνει η, το Κοινοβουλίο και η Επιτροπή μα σε θέματα πλούστευση απλοποίηση. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω και τα μέλη τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, γιατί μου πρόκειται για θέματα κοινή αρμοδιότητα. Να καλωσορίσω εκ βάθου καρδία και τον συνάδελφο Έλλερ, ο οποίο από πλευρά τη ε, πλευράς της Επιτροπής ε, ε, Βιομηχανίας ασχολείται με τα θέματα αυτά. Σήμερα λοιπόν θα ελέγξουμε εις βάθος τα προγράμματα τα ερευνητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι και προσβλέπω στην ανταλλαγή αυτή απόψεων. Να σας πω ότι πρέπει να δείξουμε προσοχή γιατί κάθε ταμείο είναι διαφορετικό και πρέπει σε κάθε περίπτωση να βρίσκουμε λύσεις και στα ειδικά ταμεία. Έχουμε τα δυτικά ταμεία, τα αγροτικά ταμεία, το ταμείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου, το κοινωνικό ταμείο και πάρα πολλά άλλα ταμεία τα οποία πρέπει να τα εξετάσουμε εις βάθος όπως και σήμερα το απόγευμα κάνουμε για το Ταμείο έρευνά, Να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία α, για την οργάνωση της σημερινής ημερίδα και να δώσω τον λόγο κατευθείαν για να ξεκινήσουμε στον πρόεδρο Αρτουή. Εγώ προτείνω να είστε εσείς πρόεδρος αυτής της πρώτης, αυτού του πρώτου τμήματος της συνεδρίασής μας. Μάλιστα και να δώσω την το λόγο κατευθείαν στον κύριο Βαλμπρόκ, ε, διευθυντή ε, των θεμάτων ε, γενικών υπηρεσιών. Συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια και σε θέματα απλούστευσης του προϋπολογισμού έχουμε πετύχει διάφορα στοιχεία. Και μακάρι αυτό που πετύχαμε ε, για το προπολογισμό να τα πετυχαίναμε και για όλα τα ταμεία. Και σας δίνω λοιπόν παραπάνω λόγο, κύριε Βάλμπρουκ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε σήμερα να σας κάνω μία παρουσίαση της μελλοντική πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος, ε, πράγματι πρέπει να ε, ειδωθεί στο πλαίσιο της ε, πρωτοβουλίας του προπολογισμού βασισμένη στα αποτελέσματα, που είναι μια βασική ε, φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, έχει να κάνει και με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού ε, πλαισίου. Δύο βασικοί στόχοι θα μας οδηγήσουν. Ο πρώτος είναι η αύξηση της ευελιξίας ε, και ο δεύτερος είναι η αύξηση της απλοποίησης. Ο στόχος μας είναι με τους δύο αυτούς βασικούς στόχους ευελιξία και απλοποίηση θα βελτιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο της ε, εφαρμογή του προϋπολογισμού στο τμήμα του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε έρθει σε επαφή με τις εκτελεστικές υπηρεσίες, με τις ε, υπηρεσίες γενικότερα. Ήρθαμε σε επαφή και με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς σε σε μια διαδικασία ευαισθητοποίησης που έγινε στις 6 Απριλίου 2016 και τα αποτελέσματα θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω πολύ σύντομα σήμερα. Η φιλοδοξία μας είναι όχι μόνο να υπάρξει διαβούλευση, αλλά ένας πραγματικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς και γι' αυτό τον Οκτώβριο θα υπάρξει μια εκδήλωση ανατροφοδότησης με τους εμπλεκόμενους φορείς όπου θα μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε πώς λάβαμε υπόψη τις ανησυχίες τους. Ο στόχο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού θα έχει μια συγκεκριμένη μορφή. Θα ε, συμπεριλάβει όχι μόνο ε, την πρόταση αναθεώρησης του, αλλά και στοχευμένες αλλαγές για, για ορισμένα τμήματα της νομοθεσίας ε, με σκοπό να καλύψουμε τα προβλήματα της συμφόρηση που υπάρχουν σε κάποιες νομοθετικές πράξεις. Να περάσουμε τώρα στα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Ε, κάτι που δεν μας προκαλεί έκπληξη. Ε, απάντησαν βασικά οι μη κυβερνητικέ ε, οργανισμοί, οι ερευνητικοί οργανισμοί, οι ιδιώτες και εθνικές αρχές. Επίσης, όπως βλέπετε και εσείς, τα πορίσματα χωρίζονται στις γνωστές κατηγορίες, βασικά επιδοτήσεις, οι προμήθειες και επίση έμεση διαχείριση και ε, άλλα ε, οικονομικά μέσα. Βλέπετε τα διάφορα προγράμματα τα οποία αναφέρθηκαν, ορίζον 2020, προγράμματα εξωτερικής δράσης, ε, ταμεία επενδυτικά και διαρθρωτικά, Erasmus+, Κόσμε κλπ. Ποια είναι τα αποτελέσματα τώρα της δημόσιας διαβούλευσης. Είναι σαφέστατο, υπάρχει ε, ανάγκη και έκκληση ε, για απλούστευση και ακόμη μεγαλύτερη έκκληση για ευελιξία. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία θέσαμε στους εμπλεκόμενους φορείς. Θα ήθελα τώρα να εξετάσω λεπτομερέστερα τον τρόπο με τον οποίο απάντησαν στα ερωτήματα αυτά. Επίσης καθόλου περίεργο όσον αφορά τη σαφήνεια των κανόνων δεν είναι ικανοποιημένη με την κατάσταση. Ε, ζητούν ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, στο οποίο θα αναφέρονται όλοι οι σχετικοί κανόνες. Ένα επίσης ε, πολύ σαφές αποτέλεσμα, ε, πολύ μεγάλη ζήτηση στον τομέα της σύγκρουσης συμφερόντων που καλύπτει ε, κάθε ε, τρόπο εφαρμογής. Αυτό δεν αφορά ε, μόνο δικό μας, αντικιά μας ανησυχία, αλλά αφορά και την κοινή διαχείριση, αλλά και την έμεση διαχείριση. Όσον αφορά την ευελιξία, Υπάρχει έντονη υποστήριξη για τη χρήση των καταπιστευμάτων, ε, ακόμη και σε εσωτερικές κρίσεις, ε, μικρότερα αποθέματα σε ε, μηχανισμούς χρηματοδότησης για τις εξωτερικές δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει τις ανησυχίες που αναφέρθηκαν σε σχέση με την προσθετικότητα, συμπληρωματικότητα, τον καλύτερο συντονισμό, όπως επίσης και την αναζήτηση ενός κοινού συνόλου κανόνων με άλλους ε, δωρητές. Περνούμε τότε λογικά και στην επόμενη ερώτηση που αφορά την ε, αυξημένη σύγκληση κανόνων. Εδώ βλέπουμε ε, ότι ε, όσοι απάντησαν ε, ζήτησαν ε, ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, ειδικότερα όταν γίνεται συνδυασμός διαφόρων μέσων ή διαφόρων ειδών παρέμβασης. Ζητήθηκε λοιπόν διαλειτουργικότητα μεταξύ οικονομικών μέσων μεγαλύτερης σύγκλησης, έμεσης ε, διαχείρισης και επιδοτήσεων και να ε, μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο ε, οι μη συντονισμένε προδιαγραφές των διαφόρων προγραμμάτων. Κάτι ακόμη είναι τα απλοποιημένα έντυπα της εξόφλησης του κόστους. Η κατάσταση είναι λιγότερο σαφής βέβαια εδώ ε, Ε, κατά πόσο δηλαδή θεωρήσαμε, θεωρήθηκε ότι η εν μέρη πλήρης κάλυψη του κόστους ε, έχει βελτιώσει την ασφάλεια ε, δικαίου. Η ερευνητική κοινότητα και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι ακόμη πολύ επιφυλακτικοί ως προς το σύστημα εξόφλησης βάσει των αποτελεσμάτων, γιατί πιστεύουν ότι αυτό δεν θα δώσει τη δυνατότητα κάλυψης του πραγματικού κόστους και επίσης γιατί πιστεύουν ότι αυτή η νέα προσέγγιση προσέγγιση πρέπει να δοκιμαστεί πριν προταθεί. Αφού όμως ε, λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα ύπαρξης μιας εναλλακτικής επιλογής και όχι κανόνα, τότε ε, είναι κάπως πιο ε, θετική ως προς τη δυνατότητα αυτή. Αυτό που θα ήθελα επίσης να πω εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι για μας η χρηματοδότηση της έρευνας δεν αφορά ένα συγκεκριμένο μέσο, είναι ένα συνδυασμός μέσων κατά ε, ποσά, ε, επιδοτήσεις για ένα τμήμα της έρευνας, ε, άλλο τμήμα όταν πλησιάζουμε προς το τέλος του ερευνητικού προγράμματος. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρξει μια διαφορά μεταξύ ε, του, των αποτελεσμάτων βάση output και των αποτελεσμάτων βάση αποτελεσμάτων. Ε, το ένα έχει να κάνει με το παραδοτέο προϊόν που μπορεί να είναι μια δημοσίευση άρθρων, ε, συμμετοχή σε συνέδρια, ανάλυση εργαστηριακή, πολύ συγκεκριμένα πράγματα που δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου ε, και που θα έδιναν την δυνατότητα να ξεφύγουμε από το να ε, πρέπει να εξετάζουμε τους λογαριασμούς ε, και τους ε, ισολογισμούς με πάρα πολύ λεπτομέρεια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πιο πολύ εστιάζουμε στο input και λιγότερο στο output. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και σε μερικούς άλλους τομείς ε, ανησυχιών ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απλοποίηση των σχέσεων με τους διεθνείς οργανισμούς. Όλοι οι διεθνοί μας εταίροι μας ζήτησαν ε, να απλοποιήσουμε και να εναρμονίσουμε την υποβολή εκθέσεων, ειδικότερα στο πλαίσιο των υβριδικών δράσεων, δηλαδή στον τομέα της έμεσης διαχείρισης και οι περισσότεροι μας ζήτησαν να χρησιμοποιούμε περισσότερο και τις δικές τους ε, μεθόδους. Αυτή τη στιγμή βέβαια έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την έμεση διαχείριση και πάλι, αλλά για όλους τους κατηγορίες ερωτηθέντων, ε, ζητούν ε, μείωση των πολλαπλών επιπέδων ελέγχου, να υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής αξιοπιστίας. Αυτή τη στιγμή κάτι έχει γίνει αποδεκτό και έχει αξιολογηθεί και βέβαια αν γίνονται έλεγχοι για τα, για τα ε, ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει επίσης μια πάρα πολύ αυστηρή προσέγγιση από πλευράς μας, ε, ειδικότερα εφόσον οι διεθνείς εταίροι πηγαίνουν προς μια πλήρη κάλυψη κόστους ε, και η ημερομηνία D-3 για την σύναψη σύμβασης επίσης θεωρείται πάρα πολύ περιοριστική. Όσον αφορά τους απλοποιημένους κανόνες για τα ε, οικονομικά ε, μέσα, ε, ζητήθηκε πολύ έντονα μεγαλύτερη συντονισμός μεταξύ των οικονομικών μέσων και άλλων μορφών υποστήριξης, ώστε έπανεις ροές να μπορούν να επιστρέψουν στο μέσο το, από το οποίο προέκυψε το προϊόν, κάτι το οποίο θα ε, σημαίνει ότι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου στον ετήσιο προϋπολογισμό το ποσό αυτό. Και ε, ολοκληρώνοντας, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στους, στις, στους επτά τομείς επί των οποίων εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε, ως αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης για τους δικαιούχους και τους αποδέκτες ε, απλοποίηση και απλοποιημένες, ε, απλοποιημένα έντυπα για τις επιδοτήσεις, όπως επίσης και για τα καταποκοπήν ποσά. Ε, δεύτερον, από τα πολλαπλά επίπεδα ελέγχων να υπάρχει πολλαπλή ένας έλεγχος πιο οριζόντιος, ειδικότερα ε, και μεγαλύτερη εναρμόνιση των ε, ετοιμάτων υποβολής εκθέσεων, ε, επίσης πιο ευέλικτος προϋπολογισμός, πιο αποτελεσματική χρήση των οικονομικών μέσων, εστίαση στα αποτελέσματα ε, και ευθυγράμμιση της υποβολής εκθέσεων ε, σε δύο βασικές χρονικές στιγμές, τη στιγμή ε, της κατάρτισης του προϋπολογισμού και τη στιγμή του ελέγχου των λογαριασμών και μία απλούστερη και πιο λιτή ευρωπαϊκή διοίκηση. Αυτά κύριε Πρόεδρε, αυτές ε, είναι, αυτή είναι η τομή σου επί των οποίων εργάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Μπορούμε το Σεπτέμβριο να το ξανασυζητήσουμε για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε ε, μέχρι τις, την 1η Ιανουαρίου 2017, κάτι το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να επηρεάσουμε το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και Ελπίζω να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια συζήτησή μας με τους ε, πλεκόμενους φορείς για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Σα ευχαριστώ. Τα πράγματα που μα είπατε δεν είναι εντελώ χωρί αντιφάσει σε ό,τι αφορά τι διαβουλεύσει των ενδιαφερομένων μερών. Γι' αυτό λοιπόν και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα υποβάλει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι από τα βιασικά στοιχεία στο θέμα του ελέγχου, ένα από του βασικού φορεί, μάλλον, είναι το λεκτικό συνέδριο. Ε, καλωσορίζω τον κύριο Λαζάρου, ο οποίο Ε, θα μα μιλήσει εξ ονόματο του λεκτικού Συνεδρίου για όσο χρειάζεται να γίνει. Έχετε το λόγο, κύριε Λαζάρου. Ευχαριστώ. Κυρία Γκρέσλε, κύριε Αρτουρί, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Ο δημοσιονομικός κανονισμός θέτει το πλαίσιο για την χρηστή χρηματοδοτική διαχείριση των ευρωπαϊκών πιστώσεων πρέπει να δαπανώνται οι πιστώσεις αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υπάρχει έλεγχος ε, με διαφάνεια για τον τρόπο αυτό. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω κάποιες προσωπικές απόψεις. Ο προηγούμενος ομιλητής μας έδωσε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις προβλέψεις της. Σύμφωνα με τη συνθήκη, εμείς θα γνωμοδοτήσουμε επ' αυτόν, αυτή τη οι προτάσεις αυτές είναι διαθέσιμες και σε έφετο χρόνο πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σήμερα μπορούμε όμως να σκεφτούμε το πώς θα είναι ο δημοσιονομικός αυτός κανονισμός και πώς μπορεί να βελτιωθεί μέσω βελτίωσης κάποιων πρακτικών θεμάτων που προέρχονται από την καθημερινή μας εμπειρία. Θα ξεκινήσω με κάποιες γενικές παρατηρήσεις επί των αρχών και μετά θα έλθω σε θέματα κάπως πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η χρηστή πρακτική δεν προαπαιτεί αυστηρές ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα όργανα πρέπει να διαχειρίζονται τις δαπάνες αυτές με νόμιμο και τακτικό τρόπο. Οι δράσει της διαχείρισης είναι το κλειδί της βελτίωσης αυτής της διαδικασίας. Οι δαπάνες αυτές δεν θα πρέπει να γίνονται με καταχρηστικό τρόπο και θα πρέπει να παράγουν τα βέλτιστα αποτελέσματα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Απαιτείται λοιπόν έγκαιρη και διαφανής διαδικασία ελέγχου. Ε, το δημοσιο... Ο δημοσιονομικός κανονισμός θέτει το πλαίσιο για τη χραστή διαχείριση, ποιος κάνει, τι κάνει, πότε το κάνει και πώς το κάνει. Νομίζω ότι το τελευταίο κομμάτι, ο έλεγχος και οι ευθύνε για αυτά τα οποία έχουν γίνει ενδιαφέρουν το ελεγκτικό συνέδριο. Και ε, θα μπορούσα να σας δώσω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για τον τρόπο που κάνουμε. Είμαστε στην τελική φάση ε, διαβούλευσης ε, και συμβουλών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Είμαι μέλος σε αυτήν την ομάδα η οποία θα δημοσιεύσει την έκθεσή της στο φθινόπωρο. Το θέμα του υπολόγου είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της προσπάθειας και θα φαίνεται καλύτερα στον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωθεί στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης ο δημοσιονομικός κανονισμός. Ε, στην συνάντηση την οποία είχε οργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2016, όπως είχε πει και ο πρόεδρος Αρτουή, e, ε, η κοινή λογική πρέπει να μας καθοδηγήσει. Αυτό εγώ το ερμηνεύω σαν την επιλογή και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Δηλαδή, συμμόρφωση ή εξήγηση στην περίπτωση απόκλησης. Νομίζω ότι το εσωτερικό ε, δίκτυο ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλες σεβαστές υπηρεσίες παίζουν και αυτές τον ρόλο τους. Υπάρχουν βέβαια σημεία τα οποία υπογραμμίσαμε στο παρελθόν και παραμένουν. Θα πρέπει για μια ακόμη φορά ε, οι επιπλέον υποχρεώσεις να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο κατά τη διάρκεια αυτής της πολιετούς δημοσιονομικής περίοδου δημιουργούν προβλήματα σε σχέση με τις υπερβολικές δαπάνες εξυπηρετούν τον στόχο του σωστού προγραμματισμού των πληρωμών τα δημοσιονομικά μας μέσα παρακολουθούνται σωστά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εγκαίρως και μπορεί να τις δώσει ε, στην φάση που απαιτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε σχέση με τα έσοδα Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες για την αντιμετώπιση υψηλών ισοών. Σαν παράδειγμα στην γεωργία ο προϋπολογισμός για άμεση βοήθεια προς τους γεωργούς μειώνεται κατά αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Από τη μία θα πρέπει να προγραμματίζει κανείς την δαπάνη χονδρικά από την αρχή όπως προβλέπεται. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη βέβαια. Ο προϋπολογισμός είναι εκεί για να βοηθήσει την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δημοσιονομικός κανονισμός επιτρέπει να γίνουν κάποια βήματα στα πλαίσια ενός προϋπολογισμού ο οποίος βασίζεται στα αποτελέσματα αλλά πώς όλα αυτά θα επηρεάσουν την δημοσιονομική διαδικασία και την διαδικασία απαλλαγής της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής. ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να ασχολείται και με, τον, με την δημοσιονομική διαδικασία με βάση την επίδοση, την εφαρμογή και τον έλεγχο. Η βελτίωση της ποιότητας της δαπάνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί απλοποίηση. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο συγκεκριμένη ομάδα των επιτρόπων που ασχολείται με τον προϋπολογισμό να είναι υπόλογοι και σε σχέση με τα αποτελέσματα σε επίπεδο επιδόσεων και σε σχέση με τα αποτελέσματα ε, σε επίπεδο τακτικής εκτέλεσης. Θα περάσω τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας είναι οι προθεσμίες. Οι προθεσμίες είναι ε, αναπόδραστο συστατικό ενός δημοσιονομικού κανονισμού. Πρέπει να γίνονται εγκαίρως οι διαδικασίες. Το να δίδονται οι εκθέσεις νωρίτερα είναι απαιτητική διαδικασία βέβαια, αλλά βοηθά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιλέξει και να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Δεν υπάρχουν προθεσμίες σε όλες τις διαδικασίες, σε όλες τις φάσεις και στάδια. Παρ' όλα αυτά, η, η εκ των προτέρων υιοθέτηση σαν παράδειγμα των Earlier των ενοποιημένων λογαριασμών για το 2015. Είναι κάτι που μαζί με την ετήσια έκθεσή μας της 13ης Οκτωβρίου, ένα μήνα νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια, θα βοηθήσει την διαδικασία. Το να γίνουν όλα αυτά λίγο νωρίτερα θα επιταχύνει επίσης και τη διαδικασία απαλλαγής. Θα πρέπει όμως ε, να έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία για την απαλλαγή που είναι απαραίτητα εννοώ ε, και να συγκρίνουμε το πακέτο της απαλλαγής. Ε, δυστυχώς η πρακτική αυτή σε κάποιες άλλες προθεσμίες δεν ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση ιδιαίτερα σχετικά με την παραλαβή των δεδομένων από εθνικές αρχές. Οι προθεσμίες αυτές είναι διάσπαρτες σε επιμέρους τομεακούς κανονισμούς και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Έπρεπε να υπάρχει εναρμονισμός εδώ. Λοιπόν, ε, δεν χρειάζονται αλλαγές τα πάντα στο εσωτερικό του δημοσιονομικού κανονισμού, αλλά σωστή εφαρμογή Σαν παράδειγμα, οι διαδικασίες με υψηλά, συστηματικά υψηλά επίπεδα λάθους πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου. Το 32.5 του δημοσιονομικού κανονισμού μας δίνει αυτές τις δυνατότητες σε, μένα, σε εμάς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαιτείται λοιπόν η διαδικασία αυτή να βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και να είναι τόσο λιπτομερής όσο αυτό είναι απαιτούμενο. Θα πρέπει επίσης να στοχεύει σε μακροπρόθεσμους στόχους να προετοιμάζει για έναν προϋπολογισμό ο οποίος να έχει σαν στόχο τα αποτελέσματα, να διευκολύνει μια σωστή σχέση ελεγχομένου και ελεγκτή σε έγκαιρη ε, χρονικά διαδικασία, να κρατήσουμε ότι είναι καλό και να μην προσθέτουμε και βαρύνουμε την διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμες αυτές τι σκέψεις που μας παρουσιάσατε. Θα τι σκεφτούμε. Food for thought. Θα πρέπει να συνεχίσουμε διάφορα, να συζητήσουμε ε, διάφορα ζητήματα για το πώς θα μπορούν να εφαρμοστούν. Το θέμα της έρευνας ασφαλώς ε, μας αφορά όλους μας. Ε, γιατί εκεί βρίσκεται το μέλλον τη Ευρώπη, Στο Ταμείο λοιπόν της έρευνας. Καλωσορίζω λοιπόν από την Ένωση της Έρευνας και της Τεχνολογίας την κυρία Ατερνέ και τον κύριο Σούτνερ. Έχετε 15 λεπτά από κοινού. Δεν είναι πολλά, αλλά νομίζω ότι θα χρειαστεί και θα μπορέσετε να τα μοιράσετε μεταξύ σας προκειμένου να μας παρουσιάσετε αυτά που θέλετε, κυρία Ατερνέ. Κύριε Ατερνέ. Μια ερώτηση προ τον κύριο Λαζάρο. Στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαδικασίας είδα ότι σε σχέση με τους πόρους εξετάζουμε και το θέμα της μείωσης των δαπανών. Έτσι όπως το παρουσιάσατε εσείς, πιστεύετε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την ονοματολογία μας, τη λογιστική και τη δημοσιονομική και να μην βάζουμε κάποιους πόρους μειώνοντας τις δαπάνες, έτσι ώστε θα έχουμε μια δημοσιονομική εικόνα πιο προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα. Αυτό εννοείται. Uh, Ελπίζω να παρακολούθησα σωστά την ερώτησή σας. Εμείς δεν προτείνουμε να υπάρξει με οποιοδήποτε τρόπο κάποια μείωση των πόρων. Όπως είπαμε και στην έκθεσή μας για το 2014, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτος και να είναι επίσης σε θέση να αντιμετωπίσει απρόβλεπτα συμβάντα και γεγονότα όπως αυτά τα οποία βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο. Ταυτόχρονα ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει μεγαλύτερα επίπεδα ευελιξίας σε σχέση με τις δαπάνες αυτές και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το λάβει υπόψη. Το καταλαβαίνω, αλλά αυτό το οποίο μου έκανε κάποια εντύπωση είναι ότι σε ορισμένα τμήματα των προϋπολογισμών παίρνουμε το καθαρό της διαφοράς ανάμεσα στις δαπάνες και τους πόρους που μπορούμε να έχουμε όπως ας πούμε οι αμοιβέ των, εργα... των εργατών υπαλλήλων. Μήπως θα ήταν προτιμότερο να φαίνονται ξεχωριστά οι δαπάνες στις δαπάνες, στις στήλε των δαπανών και τα έσοδα, οι πόροι στα δημοσιονομιστή στήλε για τα έσοδα. Um, yes, we, we, we Βεβαίως, το πιστεύουμε αυτό. Σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο προτείνουμε ο προϋπολογισμός να μην μειωθεί μέσα από τη διαδικασία του assigned revenue, το οποίο θα πρέπει στο μέλλον να συλλεγεί εκ νέου. Εμείς πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες και το λεγόμενο assigned revenue θα πρέπει να συνδέεται με το σύνολο των εσόδων. Και έτσι θα μπορεί να χρησιμοποιείται στα πλαίσια ε, του συνόλου του προϋπολογισμού. Πολύ σας ευχαριστούμε. Να συνεχίσουμε με την ε, κυρία Τάνη και τον κύριο Σάτμερ. Έχει το λόγο. Πολύ σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους δύο πρόεδρους για την ε, πρόσκληση τους σήμερα. Εν συντομία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εξ ονόματος του συναδέλφου μου να μην τα κάνουμε αυτά δύο φορές. Εν συντομία, γιατί δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να μιλήσουμε με, το, με την Επιτροπή σας. Η ΕΡΤΟ λοιπόν αποτελείται από 150 μέλη και αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μας σε θέματα και της ε, ε, Επιτροπή σας, το θέμα της έρευνας είναι τα βασικά μας ε, ζητήματα. Δεν είμαστε ούτε η μηχανία, ούτε ο ακαδημαϊκός κόσμος, ούτε τα πανεπιστήμια. Είμαστε δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο τέτοιο στόχο. Οι υπηρεσίε μας είναι συμβάσει ε, ερευνητικέ προ τι κυβερνήσει, προ τον κλάδο, το βιομηχανικό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο, ο ορίζοντα 2020 αποτελεί το βασικό πλαίσιο των εργασιών μα. Έχουμε πολλά σχόλια για τον κανονισμό. Γιατί σε ό,τι αφορά τον ε, ορίζοντα 2020, αυτό αποτελεί το βασικό στοιχείο χρηματοδότησή μα. Για να σα δώσω λοιπόν, να σα δείξω συντομία το τι συζητάμε και νομίζω ότι εδώ στην Επιτροπή σα βλέπετε διάφορε προτάσει για τον προπολογισμό. Να πω το εξή λοιπόν, ότι σε κάποιε περιπτώσει, όταν εξετάζουμε τα χρηματοοικονομικά μέσα, και λέμε ότι αυτό είναι ο τρόπο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον, έχουμε αμφιβολίε για το επιχειρηματικό μα μοντέλο. Βασίζεται σε επιδοτήσει. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια μικρή έρευνα φέτο για να εξετάσουμε τα, ε, πρώτα, τα εννέα βασικά οργανώσει έρευνα και τεχνολογία. Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τον αντικτύπο της έρευνας για το μέλλον, κοιτώντα μόνο τα θέματα επιστροφής φόρων και τα θέματα τα αφορολογικά και τα οικονομικά. Κάποιες φορές λοιπόν έχουμε την αίσθηση ότι κοιτώντα τα θέματα αυτά, τα εργαλεία αυτά, τα χρηματοοικονομικά, δεν έχουμε σωστή εντύπωση. Δραστηριοποιούμαστε στον ορίζοντα 2020, φυσικά στα τα ταμεία που υπάρχει κοινή διαχείριση, αυτό δεν είναι επιτάπητος. Κοιτάμε λοιπόν με τα, τη βάση δεδομένων της ΕΚΟΝΤΑ και είδαμε ότι περίπου 8% των ε, κονδυλίων ε, του ορίζοντα 2020 ε, έχουν δοθεί σε μέλη ΕΑΡΤΟ. Και σε 42% των project δραστηριοποιούμαστε σε ό,τι αφορά τον ορίζοντα 2020. Και αυτό φυσικά επηρεάζει πάρα πολλέ από τι δραστηριότητε σε ό,τι αφορά τον ορίζοντα 2020. Να σα δώσουμε λοιπόν αυτά τα για να σα δώσουμε μια αντίληψη του τι κάνουμε περίπου. Ε, καταρτήσαμε ένα έγγραφο και έχετε λοιπόν το λόγο Βόλφκο για να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που έχουμε να μιλήσουμε μπροστά σας σήμερα γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν συμμετέχω και στην όλη διαδικασία του λόμπινγκ. Είμαι πιο πολύ από, την, από το πλαίσιο της ε, κατάρτισης της μηχανικής σε ό,τι αφορά τις ε, αλλά μιλάω τώρα σήμερα εδώ εξ ονόματο όλων των RTOs από όλη την Ευρώπη ω πρόεδρο τη Ομάδα εργασία των δημοσιονομικών εμπειρογνωμόνων στην ΕΑΡΤΟ. Θα ήθελα να τονίσω κάποια ζητήματα, κάποια ζητήματα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα σε σχέση και όλα με αυτά που είπε και ο συνάδελφο από το Ελεκτικό Συνέδριο. Θέματα τα οποία όμω είναι πάρα πολύ σημαντικά για του οργανισμού ε, έρευνα και τεχνολογία. Σε ό,τι αφορά την χρήση των οικονομικών εργαλείων κοιτώντα την έρευνα και την ανάπτυξη, τα οικονομικά εργαλεία όπω τα δάνεια δεν δουλεύουν για σημαντικέ ομάδε όπω είναι για παράδειγμα τα RTOs, οι οργανώσει έρευνα και τεχνολογία. Και γιατί. Γιατί συχνά απαγορεύεται να παίρνουν δάνεια οι φορείς αυτές από τον νόμο ή από το κρατικό τους ή το επιχειρηματικό τους μοντέλο και η οικονομική τους δομή δεν τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν τέτοια δημοσιονομικά εργαλεία για την χρηματοδότησή τους. Και αυτό είναι μία αξιολόγηση, μία εκτίμηση στην οποία έχουμε καταλήξει μετά από τα μέτρη συζητήσεις και με την ΕΤΕΠ στο παρελθόν από δική μα πλευρά. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι το εξή, ότι τα οικονομικά μέσα μπορούν να ε, είναι μόνο συμπληρωματικά προ τι επιδοτήσει, γιατί υπάρχουν τομεί όπου έχει νόημα να χρησιμοποιούνται, αλλά συμπληρωματικά, όχι να αντικαθιστούν τι επιδοτήσει. Και από την άποψη λοιπόν αυτή είναι σημαντικό τα μέσα για τα προηγμένα οικονομικά εργαλεία να μην ε, αφαιρούνται από τα προγράμματα για να μειώνουν τις επιδοτήσεις, αλλά να υπάρχει συμπληρωματικός χαρακτήρας σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση αυτή. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που μας απασχολεί. Το κατά πόσον η χρήση κατά αποκοπήν ναι, ποσών και των ε, μονάδων, ε, των κόστων μονάδας θα πρέπει να αυξηθούν. Προφανώς πρόκειται για εργαλεία απλοποίησης και εμείς εργαζόμαστε και για μικρούς και μη έμπειρους, ε, αν θέλετε, δικαιούχους, για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή τους. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αυτό παρουσιάζεται συχνά ως μία ενιαία λύση, κομμένη και ραμμένη. που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσεις, όπως και για οργανώσει, έρευνας και τεχνολογίας ή για μεγάλες επιχειρήσεις. Και ποιο είναι ο αντίκτυπο, λοιπόν. Σημαίνει ότι α, υψηλής ποιότητας και εξειδικευσής ε, υποδομές και άτομα μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα έρευνας οι απλοποιημένες μορφές ε, αποζημίωσης από ό,τι έχει φανεί δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες ε, δραστηριότητες ε, έρευνας και ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι one size fits all, ότι μπορούν να υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ενιαίες λύσεις για όλου αυτούς τους φορείς προκειμένου να είναι και λοιπόν το συμπέρασμά μας είναι ότι αυτά τα πόσα κατά αποκοπή και τα κόστη μονάδας δεν θα πρέπει να γενικευτούν. Θα πρέπει να βρίσκονται για όσους τα χρειάζονται, αλλά να μην αποτελούν τον κανόνα για όλους τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει ε, η χρηματοδότηση των πραγματικών εξόδων να συνεχιστεί και η χρηματοδότηση του πλήρους κόστους όταν αυτό προέρχεται από ένα επαγγελματικό σύστημα χρηματοδότησης ε, προγραμμάτων όπως αυτά που χρησιμοποιούν τα RTOs. Σε ό,τι αφορά την απλοποίηση του ελέγχου και της υποβολής εκθέσεων, καλωσορίζουμε την πρόθεση απλοποίησης των κανόνων προκειμένου ο έλεγχος και η υποβολή εκθέσεων να είναι πιο ε, ε, εύκολη διαδικασία. Γιατί αυτά πραγματικά επιβαρύνουν υπερβολικά σε κάποιες περιπτώσεις και κοιτώντας και τα προγράμματα έρευνας, η έλεγχη και η ερμηνεία των κανόνων θεωρείται παράγοντα κινδύνου για του δικαιούχου. Και η εμπειρία μα λοιπόν τι λέει σε όλη τα άρτια στην Ευρώπη. Λέει ότι ένα πρόβλημα είναι ότι φαίνεται να υπάρχει ένα κύκλο ζωή σε ό,τι αφορά του ελέγχου κατά τη διάρκεια του ενό προγράμματο. Γιατί μπορεί να μην αλλάξουν οι γραπτοί κανόνε, η προσέγγιση όμω ενδεχομένω αλλάζει από πλευρά του δικαιούχου σε περίπτωση που, για παράδειγμα, οι μετέπειτα έλεγχοι καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα από την πρώτη έλεγχη. Και φαίνεται ότι δεν είναι ξεκάθαρο λοιπόν το τι θα πρέπει να πετύχουν. Κάτι άλλο που βλέπουμε. Είναι ένα αντίκτυπο που αυξάνεται σε ό,τι αφορά τα αδερφωτικά ταμεία, για παράδειγμα. Ή σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης των προγραμμάτων σε άλλους ε, σε άλλες φαντότητες ε, όπως είναι ο ορίζοντας. Ε, και θα πρέπει λοιπόν, συμπεραίνουμε, να υπάρχει συνεπής και σταθερή εφαρμογή των κανόνων στους ελέγχους και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός όταν πρόκειται για μικρές ε, επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση των πόρων αυτών. Και θα ήθελα να παρουσιάσω και ένα τελευταίο σημείο. Το θέμα των ελέγχων βάσει output, βάσει αποτελέσματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζουν οι οργανώσει έρευνα και τεχνολογία. Και ξέρετε, επί τη αρχή είναι ελκυστική η ιδέα αυτή, γιατί αποτυπώνει τη δέσμευσή μα να υπάρχει τέτοιο αντίκτυπο στην ε, ενέργεια έρευνα και ανάπτυξη και τεχνολογία. Αλλά στην παρούσα φάση χρειαζόμαστε πολύ πιο πολλέ πληροφορίε και πολύ πιο πολλά στοιχεία για να ενημερωθούμε και να ξέρουμε κατά πόσον θα πρέπει να προτιμηθεί αυτή η οδό. Αυτό που είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μα είναι το εξή, ότι η έρευνα συμπεριλαμβάνει εξορισμού κίνδυνος. Το... Η μέτρηση του αποτελέσματος είναι κάτι το προβλέψιμο. Αυτή λοιπόν η αδυναμία προβλέψιμότητας ενδεχομένω να βοηθήσει τα μελλοντικά προγράμματα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο όμως εδώ πέρα συνάδουν αυτά τα δύο. Ένα από τα ερωτηματικά που έχουμε Η έννοια λοιπόν αυτή θα πρέπει να αναπτύχθει με τη συμμετοχή των βασικών ε, φορέων. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου σε τελική αναλύση να υπάρχει και αποδοχή. Και συμφωνία ότι μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό και επίση είναι σημαντικό τα διάφορα θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα στο Ελεκτικό Συνέδριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να έχουν την ίδια αντίληψη για του ελέγχου βάσει αποτελέσματο. Γιατί αυτό είναι βασικότατο για να επιτευχθεί ένα απαιτακτό επίπεδο νομική βεβαιότητα για του δικαιούχου. Αυτό λοιπόν θα συστήναμε πισταμένους και κατεπηγόντω σε ό,τι αφορά τι προσεγγίσει των ζητημάτων αυτών. Βλέπω ότι τελείωσε και ο χρόνο μου. Αυτά ήταν κάποιε συγκεκριμένε ε, σκέψει που είχα να παρουσιάσω από το ιστορικό τη ε, κοινότητα των RTOs και θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερω ε, αν λαμβάνετε υπόψη και τις δικές μας σκέψεις λοιπόν για τις μελλοντικές σας εργασίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις αυτές και απογοητεύτηκα κάπως ε, σε ό,τι αφορά την απροθυμία σας για τα καταποκοπή ποσά. Γιατί πρόκειται για το εξορισμό εργαλείο υπέρ τη απλούστευση. Καταλαβαίνουμε και το πρόβλημά σα, λοιπόν και ότι χρειάζεται όμω και νομική βεβαιότητα σε ό,τι αφορά του εκ των έλεγχους. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχει ανάγκη να ενεργήσουμε. Δεν θα είναι απλό να εκτιμήσουμε προ ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ενεργήσουμε βέβαια. Σα ευχαριστούμε για την παρουσίασή σα. Και συνεχίζουμε με τον ε, τον ε, Μετεφυρεάλης, μια γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας. Και έχετε το λόγο. Νομίζω ότι κάποιο λάθος έκανα, λέει πρόεδρος, και ξέχασα τον κύριο Έστερμαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων. Με συγχωράτε. Έχετε το λόγο members of the committee, the members of parliament. I would first like to thank you for inviting us to share the views of the European University Association. and... Για να παρουσιάσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων και πριν αρχίσω να πριν αφαιρθώ στα σημεία τα οποία εμείς θέσαμε στη δημόσια διαβούλευση. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για την ένωσή μα. Είμαστε η μεγαλύτερη ένωση πανεπιστημίων, πάνω από 800 ε, μέλη από 47 χώρε και έχουμε ε, 33 ε, ενώσεις, εθνικές ενώσεις ε, πανεπιστημίων ε, με εκπροσώπηση διαφορετικών συστημάτων στην κοινότητά μας. Εμείς υποστηρίζουμε τους διαμορφωτές πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά μέσω συντηρητικών δεδομένων, διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών όπως κάνουμε και τώρα για τη διαβούλευση για το Erasmus Plus και τον Ορίζοντα 2020. Έχουμε εργαλεία για το benchmarking όπως ένα δημόσιο παρατηρητήριο και και προσπαθούμε να δίνουμε πάντοτε μια ευρύτερη προοπτική σε συζητήσεις όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Χώρο και την ε, Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση. Επίσης, δέκα συγκεκριμένα σημεία ε, τα οποία προσπάθησαν να δουν την ευρύτερη εικόνα στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και πριν αναφερθώ σε αυτά τα δέκα ξεχωριστά σημεία. Θα ήθελα να σας πω ποια κατά την άποψή μας, κατά, την άποψή είναι οι βασικές ε, προκλήσεις ε, της βιωσιμότητας και της ευελιξίας από την πλευρά των πανεπιστημίων. Βλέπετε σε αυτήν την διαφάνεια τα δεδομένα από το, δημο, από το παρατηρητήριο δημόσιας χρηματοδότησης από το 2008 μέχρι το 2014 πολλά ε, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης έχουν μειώσει χρηματοδότηση μέχρι και 50% ε, για τα ερευνητικά προγράμματα και τα προγράμματα τα εκπαιδευτικά. Αυτό φυσικά έχει σημαντικό αντίκτυπο ε, για τα συστήματα χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη. Το πρώτο ε, σημείο το οποίο ε, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και το ακούσαμε και από ε, τους προλαλήσαντες, το να υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, είναι σημαντικό να υπάρχουν βέβαια και διάφορες μορφές χρηματοδότησης παράλληλα και διάφοροι τομείς και δικαιούχοι. Γιατί είναι μια ακόμη δυνατότητα για τον ορίζοντα 2020 και το Erasmus Plus να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες ε, της ε, ακαδημαϊκής έρευνας και εκπαίδευσης. Το δεύτερο σημείο είναι κάτι που επίσης ε, αναφέρθηκε ήδη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ του προπολογισμού βάση προ, ε, αποτελεσμάτων και της χρηματοδότησης βάσης κόστους, βάση κόστους ε, ο υπολογισμός του αντικτύπου και των αποτελεσμάτων είναι ε, μεγάλη πρόκληση, ειδικά στον ερευνητικό τομέα, είναι πολύ μεγαλύτερη πρόκληση για την βασική έρευνα. Ε, το ίδιο ισχύει και σε πολλά εθνικά συστήματα, οπότε ελπίζουμε ότι αυτό ε, επίσης θα ληφθεί υπόψη και ότι θα υπάρξει πρόσκληση προς τους εμπλεκόμενους φορείς να ε, συνεισφέρουν στην συζήτηση αυτή προσμέτρηση των αποτελεσμάτων είναι επίσης ε, πρόκληση για την βασική έρευνα, γιατί το κανένα αποτέλεσμα μπορεί και αυτό να είναι μια σημαντική ανακάλυψη και αυτό είναι μια σημαντική πτυχή συνεπώς. Για, του, για τα πανεπιστήμια είναι πολύ σημαντικό η χρηματοδότηση να βασίζεται στο κόστος της ε, δραστηριότητας, ε, ώστε να εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα και πράγματι οι μονάδες κόστους ε, για τα καταποκοπήν ποσά είναι σημαντικές πτυχές απλοποίησης, ε, α, όμως πρέπει να υπάρχει και η διασφάλιση ότι υπάρχει επαρκής κάλυψη του κόστους. Ε, και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως ακούσαμε, ως προς αυτό. Τρίτο σημείο το οποίο θα θέλαμε να επισημάνουμε αφορά τις ε, ε, διοικητικές διαδικασίες. Ε, υπήρξε σημαντική βελτίωση όσον αφορά τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την επιδότηση. Μερικές φορές όμως μπορεί να πάρει χρόνο για μεγάλες κοινοπραξίες και είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια ευελιξία. Κάτι ακόμη που θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για την ε, κάλυψη του κόστους και ο δημοσιονομικός κανονισμός το επιτρέπει αυτό. Είναι σημαντικό όμως και οι διάφοροι δικαιούχοι να μπορούν να διαλέξουν γιατί θα υπάρξουν ε, δικαιούχοι πανεπιστήμια που θα προτιμούσαν ε, μία καταποκοπήν επιλογή γιατί δεν έχουν ε, την ικανότητα οικονομικής διαχείρισης, δεν έχουν τόσα πολλά προγράμματα να διαχειριστούν και υπάρχουν άλλα ιδρύματα που έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα και θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους διαδικασίες διαχείρισης και λογιστικού ελέγχου. Πέμπτο σημείο, θα ήταν σημαντικό να βελτιώσουμε τη συμβατότητα, να βελτιώσουμε τη συμβατότητα των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο εμείς από διαβούλευση με τα μέλη μας βλέπουμε ότι η συγχρηματοδότηση, η αρχή της συγχρηματοδότησης ε, αποτελεί μια πρόκληση. Μπορώ να σας δώσω μερικά ε, παραδείγματα. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν, υπάρχει συγχρηματοδότηση, το υπόλοιπο τμήμα ε, προέρχεται κατά 80% από το βασικό προπολογισμό. Οπότε όσοι έχουν αρκετή χρηματοδότηση μπορούν να, να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα Όσοι όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα, αντιμετωπίζουν και πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, ε, ειδικά σε εθνικό επίπεδο. Η εθνική και η περιφερειακή διάσταση λοιπόν ε, θα ήταν ε, ένας, ένας καλός τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Έκτο σημείο που προέκυψε στη διαβούλευσή μας είναι η αποδοχή των εθνικών πρακτικών διαχείρισης και ελέγχου αυτό θα έπρεπε να εφαρμόζεται περισσότερο, γιατί θα ήταν ένα από τα βασικά ε, στοιχεία που θα συνέβαλαν στη μείωση του διοικητικού άχθους και στην απλοποίηση και θα οδηγούσαν τελικά σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Δύο τρίτα ε, των πανεπιστημίων ε, πρέπει να οργανώσουν παράλληλες διαδικασίες ελέγχου για, το, για τον ορίζοντα 2020 αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά χρήματα ε, σπαταλώνται κατά αυτόν τον τρόπο. Σημείο 7 είναι η ελπίδα ανάπτυξη ε, μιας προσέγγισης βασισμένη στην εμπιστοσύνη προς τους δικαιούχους όσον αφορά τι διαδικασίε ελέγχου, πρέπει να ε, φεύγεται ο διπλό έλεγχο και αν είναι δυνατόν να είναι αποδεκτά τα εθνικά πιστοποιητικά ελέγχου. Σημείο 8. Ελπίζουμε επίσης ότι στις περαιτέρω, στην περαιτέρω ανάπτυξη κανόνων θα υπάρξει εξισορρόπηση μεταξύ της ε, σταθερότητας των κανόνων και της ευελιξίας αυτών. Σημείο 9. Κάτι το οποίο έχουμε και πάλι ήδη ακούσει μας απασχολεί η επέκταση των νέων χρηματοδοτικών μέσων, των δανείων. Πέρσι, για παράδειγμα, ε, χρήματα αφαιρέθηκαν από τον ορίζοντα 2020 και μεταφέρθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις. Μας ανησυχεί αυτό γιατί αυτά είναι χρήματα τα οποία ε, μεταφέρονται από ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που βασίζεται σε επιδοτήσεις σε ένα άλλο πρόγραμμα και ε, ένα μεγάλο ε, ε, τμήμα των πανεπιστημίων δεν μπορούν να επωφεληθούν από ένα πρόγραμμα δανειοδότησης γιατί δεν δικαιούνται να λάβουν δάνεια ή όπως είπα όπου έχουν γίνει περικοπές δημόσιας, δημόσιων δαπανών τα πανεπιστήμια ακόμη και αν έχουν τη δυνατότητα δεν θα χρηματοδοτούν ε, αβέβαιη έρευνα ε, και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα της εφαρμογής, ε, να δουλέψει το σύστημα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό. Ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο και οι επιτροπές θα ε, δουν τις επίσημες, εξετάσουν τις επίσημες διαδικασίες και πώς μπορούν στην πράξη να λειτουργήσουν ε, οι αρχές που ε, συζητήσαμε. Αυτά ήθελα να σας πω. Είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τις διάφορες πτυχές στο νηστό τοπό μας και με πολύ χαρά να τις μοιραστούμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ. για την παρουσίαση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Και τώρα ο, ο, ο καθηγητής Φύρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας αγαπητοί πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και πάλι που μας προσκαλέσατε για την ε, εκπροσώπηση και μικρό μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια μικρή επιχειρήση. Ε, είμαστε, έχουμε έδρα στο στην Γαλλία, στα σύνορα με την Ελβετία, την Βασιλεία και την, το Φράιμπουργκ από πλευρά της Γερμανίας. Είμαστε πραγματικά μια μικρή ε, επιχείρηση η οποία εργάζεται επί των για την ε, ανάπτυξη βιολογικών δίκτων και τα προγράμματα μας, τα προϊόντα μας είναι καινοτομικά. Εξελισσόμαστε και δραστηριοποιούμαστε σε τρεις βαθικές παθολογίες που έχουν βασική αντικτύπω στην Ευρώπη. Καρδιακή ανεπάρκεια, καταρχάς, που προκαλείται από μυοκάρδιο ε, του μυοκαρδίου. Ε, για το ε, Alzheimer εργαζόμαστε επί της πρόγνωσης και της ε, έγκαιρης διάγνωσης του Alzheimer με τη χρήση κυτάρων του αίματος. Εξετάζουμε λοιπόν το αίμα και για τη ρευματοειδή ανθρίτιδα αναπτύγουμε νέες τεχνολογίες για να αξιολογήσουμε τις διάφορες θεραπείες. Γιατί είναι πολλές οι θεραπείες που διατίθενται για την ασθένεια αυτή και είναι πολύ μεγάλη η επιλογή για τον ασθενή. Είναι δύσκολο, δεν επιλέξει ο ασθενής. Άρα, σήμερα λοιπόν συναποτελούμε στα 70 άτομα ε, κυρίως στο Νίγκ, λοιπόν βρισκόμαστε, αλλά και στο Παρίσι και στο Στρασβούργο, με πιο πολλοί από εμά. Πολλά από τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρεία μας είναι από τον ακαδημαϊκό κόσμο, από τα πανεπιστήμια και έχουν ε, περάσει πολλά χρόνια σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείε. Όπως ξέρετε, στα πέριξη της Βασιλείας είναι πολλές οι φαρμακοβιομηχανίες. Και έχουμε και την κοιλάδα των βιολογικών αυτών επιχειρήσεων στη Αλσατία. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στη, στα επιλεγμένα, στις επιλεγμένες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που καταφέραμε να πετύχουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα και είμαστε πολύ περήφανοι ως Ευρωπαίοι εδώ και 5-6 χρόνια ιδιαίτερως, γιατί η εταιρεία μας είχε μόνο τρία άτομα το 2008 και υπέβαλε την πρώτο project για την ε, καινοτομική ιατρική και λάβαμε περίπου 70 εκατομμύρια χρηματοδότηση. Ε, πρόκειται για ένα μεγάλο κίνδυνο φυσικά, μεγάλο ρίσκο. Γιατί ήταν πολύ καινοτομικά τα προϊόντα τα οποία παράγαμε. Αλλά αυτό όμως καταδεικνύει επίσης πόσο αξίζει η επένδυση σε τέτοια έργα, γιατί αυτά θα χαράξουν το μέλλον. Όπως βλέπετε λοιπόν στη διαφάνεια αυτή η εταιρεία μας και οι θηγατρικές της συμμετέχουν σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα, κάποια παλαιά προγράμματα όπως το πρόγραμμα πλαίσιο, το πρόγραμμα πλαίσιο, το IMI, το πρώτο πρόγραμμα και το ορίζοντας 2020. Συμμετέχουμε επίσης και σε κάποια μικρά εθνικά προγράμματα. Και θα ήθελα να επικριθώ όμως σε αυτά τα τρία προγράμματα, τα οποία πραγματικά είναι ωφέλιμα και μας διδάσκουν πολλά. Χαίρομαι λοιπόν που σημειώθηκε και αυτή η πρόοδος τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, αλλά και την τελευταία δεκαετία. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες συνολικές εκτιμήσεις από σε μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα IMI. Και όπω βλέπατε ήταν πολύ χαμηλό ο συνολικός, ε, το συνολικό ποσοστό χρηματοδότησης αρχικά, 75%. Πλέον αυτό έχει φτάσει το 100% και νομίζω ότι τα νέα μέλη του ε, IMI2 είναι ικανοποιημένα. Τα προγράμματα του 7ου προγράμματος πλαίσια, όπως ξέρετε έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι. Υπήρχαν κάποια σημεία κριτική σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των προγραμμάτων γιατί τα αποτελέσματα αυτά κάπως ε, αποδυναμώθηκαν. Αλλά σε γενικέ γραμμέ καλή συνεργασία με αυτά συγκεκριμένα αποτελέσματα για τον ορίζοντα 2020. 9,5 στα 10 έχει πετύχει το ορίζοντα 2020. Πολύ καλή βαθμολογία. Έχουμε δύο εργαλεία για το, στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 με 5 εκατομμύρια χρηματοδότηση σε κάθε ένα από αυτά. Και φυσικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, αλλά έχει αλλάξει πάρα πολύ διαχείριση των προγραμμάτων αυτών. Για τα προγράμματα IMI είδαμε κάτι περίεργο. Ο εκπρόσωπος όλων των προγραμμάτων ε, του IMI έχω κάποιες αμφιβολίες. Αναζητήσαμε λοιπόν το τι πήγε λάθος δεν μπορέσαμε να βρούμε και τόσο πολλά στοιχεία λάθος, λανθασμένα. Άρα, αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να σας διαβιβάσουμε ως μήνυμα. Ολοκληρώθηκε ένα πρόγραμμα του IMI πέρσι και ακόμα δεν έχουμε λάβει την τελευταία δόση. Ένα χρόνο μετά την υποβολή της έκθεσης. Δεν ξέρουμε γιατί. Μήπως επειδή το πρόγραμμα αυτό του προγράμματος ε, προεδρεύει ο συντονιστής του FBI. Και ο συντονιστής αυτός δεν ε, ακολουθεί την αντιδικασία υποβολής αναφορών. Ε, δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό. είναι σημαντικό για τα προγράμματα IMI είναι, και έχουμε τρία προγράμματα IMI, ένα των οποίων έχω συστήσει και εγώ. Στο τέλος του πρώτου, του πρώτου project παρατηρήσαμε λοιπόν το εξής. το ίμιση των επιχειρήσεων του FBI δεν σεβάστηκε τις αρχικές δεσμεύσει. 16 εκατομμύρια ευρώ ε, έπρεπε να συγκεντρώσουν σε συγχρηματοδότηση 30% λιγότερη χρηματοδότηση από αυτό που είχε συμφωνηθεί. Και αυτό ασφαλώς έχει άμεση επίδραση στην υλοποίηση και στα αποτελέσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μέλη της, του FBI και επιχειρήσεις να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για την εκκίνηση των προγραμμάτων αυτών. Και τα μέλη FBI να ενσωματώνουν στους εσωτερικούς τους στόχους τα προγράμματα αυτά. Όχι μόνο να συμμετέχουν έτσι γενικά στα προγράμματα αυτά τα βασικά μας προγράμματα είναι προγράμματα ανταγωνιστικότητας. Και όλοι χρειαζόμαστε τέτοια προγράμματα και από την φαρμακοβιομηχανία, αλλά και από πλευρά των α, ε, ε, ακαδημαϊκών ε, και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να κοιτάξουμε λοιπόν τώρα το εργαλείο του ορίζοντα 2020, μου είπαν να σα δώσω ποια είναι η πρώτη εντύπωση που έχουμε και έχω σχηματίσει μετά από ένα χρόνια για το πρόγραμμα IGEA. Δεν είμαστε σε ό,τι αφορά διαγνωστική εταιρεία. Και ένα δεύτερο project. Μα εξέπληξε το πόσο εύκολη ήταν η διαχείριση των προγράμματων αυτών. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ψηφιακή διαμόρφωση των ε, χρηματοοικονομικών ζητημάτων και των διοικητικών ε, ζητημάτων. Μας ικανοποιούν και τα επιστημονικά στοιχεία και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για το πρώτο εργαλείο ε, για τις μικρομεσαίες στους κόλπους του ορίζοντα 2020 δεν σημειώθηκε καμία αναβολική καθυστέρηση. Μία, ένα στοιχείο πρόσθετης αξίας είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ε, μεγαλύτερη ε, εξουσία και μεγαλύτερη περιθώριο δράση. Φυσικά όλα αυτά προσανατολίζονται στο αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε ό,τι αφορά και τα μέλη του ομίλου. Αυτό έχει να κάνει και με τα συμβόλαια υπερβολαβίας Και φυσικά όλοι να ζητούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όλα είναι σχετικά. σεβόμαστε και άλλες τις προθεσμίας. και χάρη στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα το κόμβο, η πύλη για του ε, συμμετέχοντε, όλα αυτά μα βοήθησαν εξαιρετικά. Μα έκαναν τη ζωή πιο εύκολη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τέτοιων project. Σα ενημερώνουμε λοιπόν ότι Κατά το παρελθόν ήμασταν 6 έως 10% ε, Είχαμε 6 έως 10% ε, του συνολικού ποσού χρηματοδότηση ε, για θέματα ε, διοικητικά. Σήμερα πλέον το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο, 4-6%. Πολύ θετικό λοιπόν αυτό. Οι πρόσφατες τώρα αλλαγές για την κατάργηση επικοινωνίας μέσω χαρτιού με τα ευρωπαϊκά όργανα μας βοήθησε προκειμένου να γίνεται και πιο γρήγορα η υποβολή των αναφορών αυτών, αλλά και να υπάρχει και πιο ανοιχτή επικοινωνία. Η εισαγωγή διαρκών εργαλείων υποβολής αναφοράς άλλαξε επίσης τη ζωή μας, γιατί το χάνουμε αυτό το εργαλείο στον διακάδιο και ένα χρόνο και πλέον μας βοηθάει να παρακολουθούμε όλες τις δραστηριότητε, να σεβόμαστε όλες τις προθεσμίες και όλα τα ορόσημα. Και τώρα επικεντρωνόμαστε όλο και πιο πολύ στο σκέλος της ε, καινοτομίας και όχι τόσο στην υποβολή εκθέσεων και στην ε, χαρτούρα. Και μετά από ένα εκατομμύριο δαπάνες ε, δεν είχαμε έλεγχο Έκπληξη μου προκάλεσε αυτό, πραγματική αλλαγή. Αλλά φυσικά ευπρόσδεκτη. Και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Μειώθηκαν σημαντικά τα έξοδα διαχείρισης, αλλά και ο χρόνος που δαπανούμε για την υποβολή τέτοιων εκθέσεων. Κάθε χρόνο είναι υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων και ήταν πολύ ευπρόσδεκτη η κατάργηση κάποιων των ελέγχων. Να ευχαριστήσω λοιπόν εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αναφέρω ότι από την ίδρυση της εταιρεία μας το 2008 εισαγαγάμε μια ενσωματωμένη πλατφόρμα για τους βιολογικούς δείκτες τυφυράλης και καταφέραμε να οικοδομήσουμε ένα μεγάλο δίκτυο ακαδημαϊκών με κέντρα αριστείας αλλά και με μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Και χάρη στις σχέσεις αυτές που οικοδομήσαμε, καταφέραμε να κινηθούμε γρήγορα. Χάνουμε λιγότερο χρόνο και πλέον παράγουμε καινοτόμα τέτοια στοιχεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η κυρία Γκρέσλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και έτσι μας βοηθήσατε σε ό,τι αφορά τέτοια θέματα βελτίωσης ε, της διαχείρισης των προγραμμάτων. Χαιρόμαστε και σας ευχαριστούμε. Να δώσω το λόγο τώρα στον καθηγητή από την ε, από το Ίδρυμα Max Planck. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Η προσπάθεια απλοποίησης των δημοσιονομικών κανονισμών είναι μια πολύ σωστή προσπάθεια και πρέπει να υποστηριχθεί. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ευτυχής θα έλεγα που ήρθα σήμερα να συζητήσω μαζί σας. Σχετικά τώρα για το Ίδρυμα Max Planck. Βλέπετε εδώ έναν κύριο ο οποίος έδεσε το όνομά του, ο οποίος κάποτε είχε πει κάτι το ιδιαίτερα έξυπνο θα έλεγε. Πριν από την εφαρμογή πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη περίσκεψη. Αυτός είναι και στόχος του Ιδρύματος Max Planck σήμερα. Είναι η διάδοχος ε, κατάσταση του Ινστιτούτου Kaiser Wilhelm, το οποίο έχει ζωή άνω των 100 ετών. Είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, αλλά και ταυτόχρονα να είμαστε ανοιχτοί σε τομείς όπως η εκπαίδευση. Εδώ βλέπετε ότι ε, ωφελούμεθα τα μάλα από τον προϋπολογισμό της έρευνας ε, με 2.000 προγράμματα και 900 εκατομμύρια από το 1995 και μετά. Προσπαθήσαμε για σήμερα να σας δώσουμε κάποια στοιχεία κλειδί θα έλεγα σύμφωνα με την αρχή KISS, δηλαδή uh, Keep it simple and short. Θα ξεκινήσω με, το, uh, uh, με τα, τις δαπάνες. Εμείς είμαστε πάντα υπέρ της ε, καταποκοπήν κάλυψης των δαπανών αυτών, ελαφρύνει τη γραφειοκρατική διαδικασία, ε, καθιστά διαφανή την ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκολύνει τον έλεγχο. Δεν είμαστε σε δυνατότητα βέβαια να καλύψουμε πλήρως τα κόστη μας, τα επιπλέον, και γι' αυτό το πραγματικό κόστος κάλυψης έμεσα μέσω των καταποκοπήν επιδοτήσεων είναι γύρω στο 50% και για το Horizon 2020 είναι ίσως και λίγο πιο χαμηλό. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής και εμείς πιστεύουμε ότι το Horizon 2020 είναι ιδιαίτερος περίπλοκο και έχει πάρα πολλά μέσα ως Θα πρέπει να υπάρξει ένα πιο, ε, με καλύτερες επιδόσεις συμπτυγμένο μέσο. Ιδιαίτερα οι δανειοδοτικές δραστηριότητες και τέτοιου είδους χρηματοδοτικά μέσα δεν ανήκουν εδώ και δεν πρέπει να εντατικοποιηθούν. Εμείς ε, χρηματοδοτούμεθα από το, δημόσιο, από το στην Γερμανία και σύμφωνα με το γερμανικό νόμο απαγορεύεται να παίρνουμε δάνεια. Ως εκ τούτου ε, ο κανονισμός μας δημιουργεί πρόβλημα. Δεύτερον, και εδώ θα υποστηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Σούτνερ, τα δάνεια για τέτοιου είδους ερευνητικές δραστηριότητες ίσως ε, να οδηγήσουν στο μέλλον ε, στην δημιουργία ε, μια στρατηγική τροχοπέδης που θα πνίξει την έρευνα. Ιδιαίτερα στην βασική έρευνα τα αποτελέσματα δεν είναι απλά μια ανακάλυψη η οποία δημοσιεύεται, αλλά είναι κάτι το οποίο βγαίνει και εμφανίζεται σε μια βιομηχανική δραστηριότητα ίσως και κάπου αλλού. Πώς είναι δυνατόν όταν τα κέρδη εμφανίζονται αλλού να καλείται η ερευνητική μονάδα να επιστρέψει τα χρήματα μετά τη δανειοδότηση. Και γι' αυτό λοιπόν δεν είμαστε υπέρ της εντατικοποίησης της δανειοδότησης και παρόμοιων μέσων. Ταυτόχρονα έχουμε ζητήσει όπως υπόθηκε ακόμα να μην υπάρχουν μεταφορές στους προϋπολογισμούς. Ε, έτσι και αλλιώ το δημοσιονομικό χρονικό περιθώριο που έχουμε είναι περιορισμένο ε, και το ποσοστό επιτυχίας μερικές φορές είναι πάρα πολύ χαμηλό, 3 με 7% και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι καλούνται να κάνουν οι ερευνητές ε, αν πετύχουν την προσπάθειά τους. Θα ήθελα επίσης ε, να έρθω στον πυρήνα της συζήτησής σας, δηλαδή πρέπει να υπάρξει μείωση της περιπλοκότητας του δημοσιονομικού κανονισμού, λιγότεροι κανόνες, μεγαλύτερη διαφάνεια, πάντα με βάση την αρχή KISS. Keep it simple and short. Και εδώ έρχεται αν θέλετε και η πρόκληση στην παρέμβασή μου σήμερα η δήλωση αυτή ίσως να προκαλέσει κάποιες συζητήσεις ανάμεσά σας για το τι σημαίνει το λεγόμενο output-based funding, η χρηματοδότηση output-based. Ε, ε, γιατί το λέω αυτό και με τόσο έντονο τρόπο, με μια ταφόπλακα. Γιατί μια πραγματικά σημαντική καινοτομία είναι αποτέλεσμα ε, μιας περιέργειας και μιας αν θέλετε εσωστρεφούς μορφής έρευνας και χαρακτηριστικό αυτής της έρευνας είναι το απρόβλεπτον του αποτελέσματός της, δηλαδή η χρηματοδότηση output-based επί τη βάση της πρόβλεψης της, του αποτελέσματος της ερευνητικής διαδικασίας ουσιαστικά κινδυνεύει να σκοτώσει την βασική έρευνα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε εμείς, αυτό το οποίο θέλουμε να ενθαρρύνουμε είναι να γίνει μια συζήτηση γι' αυτό. Α, το να εφαρμόζει κανείς μόνο αυτά τα οποία ξέρει σαν ερευνητή σημαίνει ότι θα μειώσει τις δυνατότητες που έχει. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό και υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην ιστορία της έρευνας. Ξέρετε όλη την ιστορία των τρανζίστορς. Το τρανζίστορ είναι αποτέλεσμα πέντε διαφορετικών βασικών αποτελεσμάτων, μάλλον αποτελεσμάτων βασικής έρευνας σε πέντε δεκαετίες το καθένα από τα αποτελέσματα αυτά από μόνο του ή το απολύτως άχρηστο και μόνο συνδυαστικά μπόρεσαν να οδηγήσουν σε κάτι το χρήσιμο. Ως εκ τούτου παρακαλώ μην το παρακάνετε με την χρηματοδότηση output based. Λοιπόν, ε, αυτά ήταν τα σημαντικά στοιχεία τα οποία θα ήθελα να σας πω σήμερα έχετε μια πραγματική ευκαιρία. Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού σας δίνει την δυνατότητα, την ευκαιρία να απλουστεύσετε ακόμα περισσότερο τα πράγματα, κάτι το οποίο θα διευρύνει και την συμπάθεια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος δηλαδή ο δημοσιονομικός κανονισμός μπορεί να βοηθήσει στην αποδοχή από την κοινή γνώμη της Ευρώπης. Δεν μπορώ παρά να σας ενθαρρύνω προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, δέσμευση αυτή. Και ιδιαίτερα σήμερα αυτό απασχολεί πολλούς ε, και σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσουμε και την Πορτογαλία, να συγχαρούμε και την Πορτογαλία για τον χτεσινό αγώνα και για το πρωτάθλημα. Ο κ. Τσάιλτ από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνα. Να πάρει το λόγο για τι ε, ανάγκε ε, των μελλοντικών μεταρρυθμίσεων. Δεν μπορούμε να σα κατακορίσουμε ότι δεν ε, ε, έχετε έλθει, γιατί γνωρίζουμε και την εργασίες σας από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Να σας συγχαρούμε λοιπόν και για την θέση αυτή που αναλάβατε. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και έχω την ευκαιρία να αναφερθώ σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις Επιτροπές Προϋπολογισμού και Ελέγχου των Προϋπολογισμών για τη συζήτηση αυτή και γιατί προσκαλέσατε τόσο σημαντικές προσωπικότητες ε, που για πρώτη φορά ε, μας εκφράζουν την άποψή τους για το πώς μπορούμε να, να συνεργαστούμε προκειμένου να βελτιώσουμε την ε, οικονομική και δημοσιονομική μας αρχιτεκτονική είναι ένα σημείο κλειδί ε, όσον αφορά το, τη διαχείριση του προγράμματος ε, έρευνας ε, των ορίζοντα 2020, όχι μόνο γιατί έχουμε να δούμε τους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού, αλλά επειδή πλησιάζουμε και στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του συστήματος ορίζον 2020. Μόνο λοιπόν ε, να συμφωνήσω μπορώ με τα μηνύματα που ακούσαμε σήμερα ώστε να μην ε, απομακρυνθούν χρήματα από την έρευνα και την ε, καινοτομία προς άλλους σκοπούς δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρούμε απαντήσεις στα πολλά πιεστικά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Με ενθαρρύνει το θετικό μήνυμα όσον αφορά την πρόοδο που έχουμε κάνει, οι προκάτοχοί μου έχουν μάλλον κάνει όσον αφορά την απλοποίηση του ορίζοντα 2020 σε σύγκριση με ε, τα προηγούμενα ε, ε πολιετή ε, δημοσιονομικά πλαίσια. Εμείς στη Γενική Διεύθυνση ε, Έρευνας και Καινοτομίας ε, αρχίσαμε διαβούλευση με 44.000 συμμετέχοντες και τα στοιχεία που λάβαμε κινήθηκαν προς την κατεύθυνση όσων ακούσαμε από τον καθηγητή Φυράτ σήμερα θεωρούν ευπρόσδεκτο το, ευπρόσδεκτο το απλούστερο μοντέλο το οποίο έχουμε προ, προτείνει, την επίσπευση της διαδικασίας ε, ε αποδέσμευσης της ε, επιχορήγησης, δύο στάδια στους διαγωνισμούς, ε, τη χρήση των συστημάτων των λογιστικών, των δικαιούχων ως εναλλακτική επιλογή, όχι πολύ έλεγχη για παρόμοιες δραστηριότητες και πάνω απ' όλα κάτι ε, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό ε, σύστημα ε, υποβολής ε, αιτήσεων για ερευνητικά προγράμματα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, οικογένεια των ερευνητικών ιδρυμάτων. Ο Επίτροπος ε, θεώρησε μάλιστα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και προτεραιότητα μάλιστα η ευθυγράμμιση των διαδικασιών. Είναι κάτι το οποίο, επί το οποίο εργάζεται και θα ήθελα να κάνω κι εγώ μία διάκριση μεταξύ από τη μία του δημοσιονομικού κανονισμού και από την άλλη των διαφόρων κανόνων και συστημάτων εντός του ερευνητικού προγράμματος του ορίζοντα 2020 και ειδικότερα των κανόνων συμμετοχής πολλές από τις λεπτομερέστερες διατάξεις που αναφερθήκαμε, στις οποίες αναφερθήκαμε ε, σήμερα διέπονται από αυτό ακριβώς το ε, από αυτόν ακριβώς τον κανονισμό. Ε, πολλά από όλα από όσα θα θέλαμε να κάνουμε και πολλά από όσα ακούσαμε από τους συμμετέχοντες στην έρευνά μας μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του, των εφισταμένων κανόνων του ορίζοντα 2020. Ας πούμε μερικά παραδείγματα. Ανέφερα ήδη τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αμβλύνουμε, να ανακουφίσουμε κάπως το βάρος ε, ε, των ετούντων χρησιμοποιώντας ε, δύο στάδια στους διαγωνισμούς μπορούν ε, οι ετούντες ε, να δώσουν μια πολύ ευρύτερη περιγραφή του project που προτείνουν και αν επιβεβαιωθεί μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ετούντων, συμμετεχόντων μπορούν να υποβάλουν λεπτομερέστερες προτάσεις. Επίσης κανόνες για το κόστος του προσωπικού που δεν καλύπτεται από οικονομικές οικονομικές χρήσει ε, των οποίων ο έλεγχο έχει ολοκληρωθεί. Εμεί προσπαθούμε να βελτιώσουμε το πόρταλ των συμμετεχόντων για να είναι σαφέστερα ε, τα πράγματα βάσει βέβαια των ε, στοιχείων που λαμβάνουμε από εκείνου. Εξακολουθούμε λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ δραστηριοί και δεν χρειάζεται να περιμένουμε ούτε αλλαγές στο δημοσιονομικό κανονισμό ε, ούτε στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο το οποίο θα αρχίσει να ισχύει μετά τον ορίζοντα 2020. Βλέπουμε παρόλα αυτά ευκαιρίες και στις δύο αυτές περιπτώσεις να σημειωθεί πρόοδος. Και όταν μιλούμε για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, βεβαίως συμφωνούμε με πολλές από τις ιδέες που ακούστηκαν και συνεργαζόμαστε βεβαίως με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών ε, για την βελτίωση και την απλούστευση της διαχείρισης του προϋπολογισμού μας, όπως επίσης και την ευθυγράμμιση των διοικητικών διαδικασιών και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να μοιραστούμε τις δικές μας εμπειρίες, αυτές που αποκομίσαμε κατά την απλούστευση που εμείς επιτύχαμε όταν περάσαμε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στον ορίζοντα 2020, σε συναδέλφους που διαχειρίζονται προγράμματα στη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών που σημείωσαν λιγότερη πρόοδο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα στο λίγο χρόνο που μου απομένει να αναφερθώ σε κάποιες από τις ιδέες που ακούσαμε σήμερα ε, καταρχάς, ε, το όλο ερώτημα του προπολογισμού που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα και του μηνύματος ε, της Αντιπροέδρου Γεωργίευα Βεβαίως, ε, όπως είπαν και πολλοί ε, προλαλήσαντες, ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πολύ στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων, μεταξύ των επιτροπών που συμμετέχουν στο σημερινό εργαστήριο, του ελεγκτικού συνεδρίου, των κρατών μελών μέσω του Συμβουλίου. Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε σε πιο ε, αποτελεσματικούς τρόπους και λιγότερο παρεμβατικούς για την ε, προσμέτρηση των αποτελεσμάτων, για την ποσοτικοποίηση τους. Ε, οι έλεγχοι βασιζόμενοι στο output Καταλαβαίνω ότι ως προς την έρευνα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσμετρήσει κανείς την επιτυχία ή την αποτυχία και μερικές φορές η αποτυχία ως αποτέλεσμα είναι μερικές φορές μια σημαντική επιτυχία για να προχωρήσουμε. Και πρέπει βεβαίως να το λάβουμε αυτό υπόψη. Επίσης, όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, ε, επειδή εγώ μόλις πρόσφατα ανέλαβα καθήκοντα, ε, μου έκανε εντύπωση ο αριθμός των φακέλων που υπάρχουν στο γραφείο μου, πάρα πολύ καλή ερευνητική εργασία, ε, κάπως επηρεάστηκε παρόλα αυτά από κακή αρχιοθέτηση και από ε, καθυστέρηση χρονική, ε, είτε προσπαθούμε να ανακτήσουμε τεράστια ποσά από οργανισμούς πολύ επιτυχείς και μεγάλου κύρους, ε, γιατί γιατί επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ σε αυτά τα time sheets και γι' αυτό ακριβώς πρέπει από κοινού να βρούμε έναν τρόπο ε, υπολογισμού των αποτελεσμάτων που ξεφεύγει από αυτή την παγίδα επιτυχίας-αποτυχίας. Αυτό μου κάνει και εμένα πολύ εντύπωση. Και να σας πω και μια εμπειρία που είχα πριν από μερικές εβδομάδες. Εγώ ανέλαβα στις 16 Απριλίου καθήκοντα. Στις 17 Απριλίου ήρθαν συνάδελφοι στο γραφείο μου και μου έδωσαν ένα έγγραφο 600 σελίδων που είναι η συμφωνία ε, για τις επιδοτήσεις ε, με σημειώσεις, που είναι η βάση για τον ορίζοντα 2020, ε, καλύπτει τα πάντα Ελπίζω ότι θα το αναθεωρήσουμε αυτό το γκώδες έγγραφο ε, σύντομα, ενδεχομένω να φτάσουμε σε πρώτη φάση σε ένα έγγραφο 200 μόνο σελίδων. Ε, Ευχαρίστω ε, να ακούσω και τις δικές σας αναζωογονητικές ιδέες. Ένας οι, λόγοι για τους οποίους έχουμε αυτούς τους κανόνες είναι επειδή τα κρατημέλη ή ε, συμμετέχοντες θέλουν σαφήνεια σε κάθε, για κάθε λεπτομέρεια, για κάθε πιθανή ε, κατάσταση που μπορεί να διανοηθεί κανείς. Οπότε ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να είναι πιο ευέλικτες οι λύσεις που θα βρούμε και να σας πω την αλήθεια, ακούγοντα κάποιες από τις παρουσιάσεις τις δικές σας σήμερα, βλέπω ότι πραγματικά θέλουμε να αγκαλιάσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε προσπάθεια έρευνας και καινοτομίας, θέλουμε ε, αριστεία, ε, θέλουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια ε, θα ήταν πάρα πολύ ευπρόσδεκτη. Άκουσα αυτά που είπατε όσον αφορά το μείγμα επιδοτήσεων και δανείων και καταλαβαίνω το επιχείρημα ότι πολύ από τους καταξιωμένους ε, συμμετέχοντές μας ε, είναι από τον ιδιωτικό τομέα όπου η δανειοδότηση είναι δύσκολο πράγμα. Παρόλα αυτά ελπίζουμε να υπάρχει ένα πλούσιο μείγμα διαφόρων μέσων που θα μας δίνει τη δυνατότητα ε, μιας ευέλικτης επιλογής αντιμετώπισης των διαφόρων προκλήσεων. Και Βεβαίως υπήρχε και μία δύσκολη συζήτηση που είχε γίνει κατά την εισαγωγή του, κατά την έναρξη ισχύω του Ταμείου για τις στρατηγικές επενδύσεις, ε, γιατί κατά τμήμα, ουσιαστικά ένα τμήμα του Ταμείου αυτού είχε σκοπό να χρηματοδοτήσει τον ορίζοντα 2020. Ήταν πολύ επιτυχές πάντως αυτό το ε, πρόγραμμα για την παραγωγή καινοτόμων επενδύσεων. Ε, τα δάνεια δίνουν κάποια μόχλευση σε σχέση με ε, το ποσό της χρηματοδότησης και νομίζω ότι αυτό θα συζητηθεί στο μέλλον. Οπότε, εν κατακλείδη, κυρία Πρόεδρε, με πολύ χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα. Εμείς στην γενική μας διεύθυνση είμαστε πάρα πολύ ενθουσιώδεις ε, ως προς τη σημείωση προόδου προς ένα πλουστευμένο σύστημα οικονομικής διαχείρισης και επίσης να μοιραστούμε την ε, εμπειρία μας ε, από τον ορίζοντα 2020 σε άλλους τομείς χρηματοδότησης Βεβαίω, ε, η αναθεώρηση δημοσιονομικού κανονισμού είναι μια καλή ευκαιρία να ε, προχωρήσουμε, αλλά δεν είναι η μοναδική ευκαιρία που θα έχουμε, να προχωρήσουμε εντό του υπάρχοντο νομοθετικού πλαισίου για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την πρόοδό μα και να συνεχίσουμε να προβληματιζόμαστε σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε στο επόμενο ε, πρόγραμμα πλαίσιο για να είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και πραγματικά το θέμα αυτό το αντιμετωπίζουμε λίγο με κάποια απογοήτευση το θέμα της απλοποίησης, γιατί η εμπειρία μας είναι ότι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ρυθμίσεις ε, ε, και χρησιμοποιούμε ε, ρυθμίσεις, υποσημειώσεις, ε, προκειμένου να είναι σαφή τα πράγματα και τελικά προκύπτει κάτι το ονομάζεται living documents, ε, ζωντανά έγγραφα. Ναι, το αντίστοιχο α, ε, διοικητικό αυτό για όλους. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Έιλερ όμω να τοποθετηθεί. Σα ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα καταρχάς εξ ονόματο τη Επιτροπή ε, Ήτρε να ευχαριστήσω και τις δύο άλλε επιτροπές για το γεγονός ότι σήμερα μας καλέσατε στην συζήτηση αυτή. Γιατί κάποια θέματα επιπτούν στο πεδίο αρμοδιότητα τη Επιτροπή ε, βιομηχανία. Να μιλήσω αγγλικά όμως. Να παρουσιάσω το, το θέμα από πλευράς output σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, του κανονισμούς. Τι σημαίνει αυτό για το πρόγραμμα. Από πλευράς ε, χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής και χρηματοδοτική. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας επανελέμενα ότι τώρα μας ε, λείπει το 3% που έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε κάτω από το 2% του ΑΕΠ. Και σε ό,τι αφορά την παγκόσμιο ανταγωνισμό, μένουμε πίσω σε σχέση με την Ασία και την ΣΥΠΑ. Είναι δράμα. Δραματική η κατάσταση. Ο συνδυασμό του... Το συνδυασμό των ε, μόνιμων περικοπών στο, στην, στην ε, χρηματοδότηση και το ότι one fits all μειώνει δραματικά το ποσοστό επιτυχίας. Μιλάμε για ποσοστό επιτυχίας χαμηλότερο του 6% και σε, θέμα, σε θέματα ε, παγκόσμιου ανταγωνισμού, αυτό το βλέπουμε και από άλλα προγράμματα εμπειρικά, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κάτω από 20% ή 15% ενδεχομένως να μην έχει ποτέ διεθνή επιτυχία, γιατί είναι πολύ ψηλό το κόστος για τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για πολλές ερευνητικέ οργανώσεις. Άρα το αποτέλεσμα. Άρα, πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχία σε σχέση με τον προπολογισμό και τίθεται το θέμα του που βρίσκεται η προστιθέμενη αξία σε ό,τι τις μεγάλες βιομηχανίες, το 125% κατά πόσον υπάρχει προσθέμενη αξία και περιθώριο κερδών. Δεύτερο θέμα. Πάντα υπήρχε αντίφαση μεταξύ των διαφόρων μοντέλων και των μοντέλων της απλοποίησης με τα ποσά κατά αποκοπή. Και αυτό τι σημαίνει. Και αυτό πάλι το λέω ουδέτερη διάθεση. Οι πρακτικές λογιστικών προτύπων είναι η εναρμόνιση των υλικών αγαθών στον κόσμο. Και έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο αγνοεί το γεγονός ότι ακόμα και οι δημόσιοι προπολογισμοί αγνοούν τις παγκόσμιες τάσεις και αυτό πρακτικά που οδηγεί στο ότι ο τομέας της έρευνας εξαρτάται ακόμα σε ό,τι αφορά επενδύσεις από τον δημόσιο κλάδο. Όπως και να το δούμε, αυτό ορίζουν οι κανόνες. Κατά τρίτον, υπάρχει και ένα διαρθωτικό ζήτημα. Καθορίζουμε πρακτικά το γεγονός ότι στην ευρωπαϊκή έρευνα έχουμε τρεις ε, διαστάσεις. Έχουμε τις εθνικές ε, πρακτικές, έχουμε τις εσωτερικές ε, λογιστικές πρακτικές των μέλων και τις λογιστικές πρακτικές που καθορίζει ο ιδιωτικός κλάδος. Και έχουμε και τον ορίζοντα 2020 με τα δικά του λογιστικά πρότυπα. Απόλυτα σε αντίθεση. Μάλλον αυτά είναι απόλυτα αντίθετα σε κάποιε περιπτώσει για του ε, συμμετέχοντε. Τα PPP, για παράδειγμα, στι συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού κλάδου. στην πράξη τα μέλη έχουν πέντε διαφορετικά λογιστικά πρότυπα στα οποία πρέπει να ανταπεξέλθουν. Αυτό και από νομική άποψης αποτελεί πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν που ανακύπτει είναι το εξή. Θα μπορούσε να είναι δυνατόν να αναφερόμαστε όχι μόνο σε λογιστικά πρότυπα και τέτοια συστήματα αναφοράς για τον ορίζοντα 2020 ή για το 1ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά και στα συνήθη εθνικά πρότυπα. Ποιο είναι ο κίνδυνο από πλευρά ελέγχου προπολογισμού και κατά πόσο θα ήταν πρακτικό ένα τέτοιο σύστημα. Γιατί δημιουργείται ένα πάρα πολύ περίπλοκο σύστημα, το οποίο δεν είναι το πλέον ευνοϊκό, κρίνουν πάρα πολλοί δικαιούχοι. Γιατί προσθέτει μία στρώση περιπλοκότητας επιπλέον των εθνικών πρωτεγραφών. Στην πράξη τώρα, το άμεσο κόστος ή διαχωρισμός του ορίζοντα 2020 βασίζεται στην αρχή ότι υπάρχει μια ακριβής διάκριση μεταξύ έμεσου και άμεσου κόστους και ότι αυτά είναι α, μεγέθη αδιαχώριστα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Η Κομισιόν στα έμεσα, στα άμεσα, στο άμεσο κόστος δεν συμπεριλαμβάνει όλο το άμεσο κόστο όπως είχε οριστεί στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Άρα ε, μιλάμε μεν για άμεσο κόστος, αλλά δεν περιλαμβάνονται αυτά που περιλαμβάνονταν αρχικά. Και αυτό ενδεχομένω να οδηγήσει σε κίνδυνο επιλεξιμότητας για πολλούς από τους συμμετέχοντες. Και είναι δύσκολο να προβλέψουμε και τελικά τι προβλήματα θα ανακύψουν. Το σύστημα ελέγχου. Τέταρτο σημείο. Όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα βάση ε, αποτελέσματος, το σύστημα ε, ελέγχου δεν αναφέρεται. Γιατί είναι διαφορετικό το επίπεδο της φιλοδοξίας και του πραγματικού οικονομικού ελέγχου. Δεν το λέω αυτό για να κατηγορήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Με το παρόν ελεγκτικό σύστημα φοβάμαι ότι μπορεί να μην αντικατοπτρίζεται ακριβώς η κατάσταση. Και μία τελευταία πλευρά. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι γίνεται μία προσπάθεια απλούστευσης από την άλλη εξαιρούμε πάρα πολλά πράγματα. Το ERT σαν παράδειγμα έχει τους δικούς του κανόνες. Και έχει δίκιο το ελεγκτικό συνέδριο όταν να παραπέμπει στην περιπλοκότητα αυτού του συστήματος. Είναι τμήμα του προϋπολογισμού αλλά εξαιρείται κιόλας. ζητούνται ξεκάθαροι κανόνες ε, λόγω της διαφορετικής φύσης της δαπάνης για την έρευνα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ειδική εξαίρεση, μετά απαιτούνται κατεξουσιοδότηση πράξης, ένα ξεχωριστό σύστημα λοιπόν, όπως και ίσως ένα μελλοντικό σύστημα για το μελλοντικό πακέτο για την έρευνα, κάτι το οποίο θα μας ξεφύγει από τον έλεγχο αλλά νομίζω ότι έθεσα το τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ε, δημοσιονομικού κανονισμού. Σας ευχαριστούμε και για τη διάρθρωση των προβλημάτων και χαίρομαι που σήμερα νομίζω ότι αναφέρουμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Μόνο το πρόβλημα για τα οικονομικά μέσα είναι καινούργιο. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε ήδη. Και αυτό το πρόβλημα τύφεται επειδή τα ζητήματα αυτά καταστούνται όλο και πιο σημαντικά. Στο θέμα των ε, συστημάτων ε, λογιστικού ελέγχου, το οποίο έθεσε ο κύριος Έλερ κατά πόσο θα, θα μπορούσε να υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο θα καθιστούσε την ε, διαχείριση των προγραμμάτων πολύ πιο εύκολα. Και εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα και αναμεγνύονται και με τις εθνικές προδιαγραφές. Τι γίνεται με τις εθνικές προδιαγραφές, μετράει το εθνικό σύστημα. Και μήπως ε, θα πρέπει να υποχωρήσει το ευρωπαϊκό σύστημα. Και είναι καλή ιδέα να αποτελούν ορόσημο, για παράδειγμα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και κατά πόσο αυτό μπορεί να επιβληθεί. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Και το λεκτικό συνέδριο ε, έθεσε ένα ενδιαφέρον θέμα για τις ε, ενιαίες προθεσμίες. Κατά πόσον αυτό είναι καν δυνατόν να ρυθμιστεί με νέο χαρακτήρα το θέμα των προθεσμίων και προς την ερευνητική κοινότητα. Έχω να απευθύνω το εξή ερώτημα. Τι γίνεται με τα πόσα κατά αποκοπή Η Επιτροπή έχει νόημα να αυξήσει ε, το όριο των ποσών καταποκοπεί για να τα καταστήσει πιο αλκυστικά. Ε, ή μήπως πιστεύετε ότι είναι τόσο περίπλοκο στην πράξη το σύστημα που δεν έχει νόημα στο θέμα των οικονομικών μέσων τώρα, των χρηματοδοτικών μέσων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα πρέπει να αλλάξετε και στο το καταστατικό σας. Για παράδειγμα το Ιδρύμα Max Planck. Πολύ εντυπωσιακό. Και θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είχατε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία για τη χρήση τέτοιων εργαλείων. Γιατί το αποκλείεται λοιπόν αυτό. Γιατί δεν μπορεί κανεί να στραφεί προ τον εθνικό νομοθέτη και να πει ότι κάτι θα πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Θα πρέπει να υπάρξει ένα εξυγχρονισμό. Και προ τον καθηγητή Φίρα, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Τι προτάσει θα είχατε να κάνετε για την απλοποίηση, για την αλλαγή. Γιατί Δικαίω είπατε ότι έχετε εργαστεί πολύ επί του status αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε και στο μέλλον αυτό. Σα ευχαριστώ και το λόγο ζήτησε και ο συνάδελφο Ντενάνο. Αλλά και φυσικά ο πρόεδρο Αρτού είναι πάρει το λόγο. Νομίζω ότι πράγματι αναφερθήκαμε και στο σύστημα της λογιστικής ενημέρωσης. Ε, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε εδώ είναι η πολλαπλότητα των συστημάτων που υπάρχει. Υπάρχει ζώνη ευρώ με συγκεκριμένους κανόνες σε σχέση με το έλλειμμα και το χρέος. Αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες καθορισμού αξιολόγησης αλλά ακόμα και επικύρωσης των λογαριασμών. Ε, υπάρχει φυσικά πολλαπλότητα γλωσσών και γι' αυτό έχουμε την διερμηνία, αλλά σε επίπεδο λογιστικό φοβάμαι ότι παραμένουμε σε μια ε, υπερβολική πολλαπλότητα, γιατί αλλιώς δεν θα πετύχουμε την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε επίπεδο επιχειρήσεων θα έλεγα ότι η λογιστική γλώσσα είναι η γλώσσα της παγκοσμιοποίησης. Αλλά στον τομέα των δημοσιονομικών τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχουμε διαφορετικούς κανόνες οι οποίοι επηρεάζονται από φορολογικούς πολλές φορές λόγους. Ε, απαιτείται λοιπόν μια ομοιογένεια σε σχέση με τους λογιστικούς κανόνες και δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες στην δημόσια και στην ιδιωτική σφαίρα. Αυτά τα οποία ανακαλύπτω εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ε, ε, εκτός κανόνων. Και αυτό δημιουργεί θέματα. Σαν παράδειγμα αυτά που κάνουμε σαν κοινοβούλια στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα. Επίσης ε, κάθε σύστημα εθνικό έχει και τους δικούς τους κανόνες αλλά και τα δικές της αρχές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και ε, θα ήθελα να ρωτήσω, κάθε γενική διεύθυνση έχει τους δικούς της κανόνες. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα κοινό με την κυρία Γκρέσλε, ξεκινήσαμε ένα πείραμα θα έλεγα και κάναμε και μια πρόκληση ενδιαφέροντος για κάποια κέντρα κατάρτισης, κατάρτισης επαγγελματικής κατάρτισης και όταν ζήτησα εγώ να δω ποια είναι τα έγγραφα τα οποία ζητούμε από τους υποψήφιους, είδα ότι ε, δεν υπάρχει μέλλον. Αν δεν υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο πραγματισμού και εμπιστοσύνης ε, και είδα ότι δύο διαφορετικές γενικές διευθύνσεις χρησιμοποιούσαν τους δικούς της κανόνες. Οπότε θα ήθελα να μάθω τι είναι αυτό που ανήκει πραγματικά στο δημοσιονομικό κανονισμό, στις 600 σελίδες και τι είναι το κομμάτι των 600 πάλι σελίδων το οποίο γέννησε κάθε γενική συνέλευση λες και οι υπάλληλοι είναι τρομοκρατημένοι και δεν παίρνουν καμία απόφαση αν δεν υπάρχει μια καταγραφή ε, θα έλεγα τυπωμένη κάπου. Λοιπόν, ε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πρέπει να τα λίγο τα πράγματα γιατί αλλιώς θα σκοτώσουμε και την καινοτομία. Επίσης αξιολόγηση εκ των προτέρων, απριόρι αξιολόγηση. Τώρα στον τομέα της έρευνας πρέπει να αποδειχθούμε ότι δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει το πράγμα. Και τέλος μία μαρτυρία σε σχέση με τις αποστολές που κάναμε σε χώρες της Μέσης Ανατολής και αναφέρομαι στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Και εδώ με ελέγχει ο κύριος Φερνάντες που είναι το παρόν. Οι διεθνείς οργανισμοί που χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά χρήματα μας είπαν ότι όλοι κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον διοικητικό φορμαλισμό δέκα έλεγχοι σε ένα χρόνο για μια οργάνωση εκεί τόπου. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι, να προχωρήσουμε. Ξέρετε πόσο κοστίζουν οι έλεγχοι, οι λογιστικοί. Δεν τα χρηματοδοτούν βέβαια αυτά τα πράγματα οι προϋπολογισμοί της Ένωσης, αλλά οι εταιρείε, οι ενώσεις, οι σύλλογοι κτλ. Μιλάμε για τρομακτικό κόστος, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η εικόνα που δίδουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καταστροφική. Για δώστε ένα δημοψήφισμα στον κόσμο με τέτοιου είδους πρακτικές, καλά δεν συνεχίζω. Καλώς. Θα μας δώσετε κάποιες απαντήσεις για την πολλαπλότητα αργότερα. Πάντως θα ήθελα να μάθω αν μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια γενική διεύθυνση που να συντονίζει τα πράγματα. Μήπως πρέπει να κάνετε ένα έλεγχο των γενικών διευθύνσεων για να δούμε τι τρέχει σε κάθε μία από αυτές. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Α, δεν ξέρω ποιος είχε ζητήσει πρώτος το λόγο. Λοιπόν, Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή, λέει ο κύριος Ντενανό, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να ακολουθηθεί από πράξεις. Υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία αναφερθήκαμε και εσείς ο ίδιος θα αναφέρατε κύριε Πρόεδρε που είναι εξόχως ανησυχητικά. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε ποια είναι τα προβλήματα στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να μας ε, λένε καλά λόγια επειδή δίδουμε χρήματα, μας κατηγορούν γιατί είναι πολύ περίπλοκες οι διαδικασίες. Και έχουμε ένα πρόβλημα ουσίας πώς εδώ μπροστά. Θα πρέπει οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται σήμερα να δώσουν αποτελέσματα. Φυσικά ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι κάτι το χρήσιμο, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί ένα εμπόδιο ε, στην δαπάνηση των συγκεκριμένων πιστώσεων. Τα χρήματα δεν πρέπει να μένουν μέσα στο δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά στα προγράμματα. Πρέπει να υπάρχουν απλοί κανόνες, εναρμονισμένοι κανόνες, ένα είδος σολφέζ, αν θέλετε, καθολικής εφαρμογής γιατί να έχουμε 15 διαφορετικά λογιστικά συστήματα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να είναι γνωστοί, ε, να έχουν διάρκεια, να μην αλλάζουν κάθε πρωί και να γίνονται σεβαστοί. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ανάγκη για έναν έλεγχο, αλλά όχι για πολλαπλούς ελέγχους, όχι για έναν πολυέλεγχο. Ε, αναφέρατε για μια οργάνωση στη Μέση Ανατολή με 10 ελέγχους μέσα σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν γίνονται τα πράγματα. Εγώ πριν 15 μέρες συναντήθηκα με τους διευθυντές ε, τριών ε, γαλλικών ερευνητικών οργανώσεων, το Ινστιτούτο Παστέρ, το ΣΕΝΕΡΕΣ και το ΙΝΣΕΡΝΑ και μας είπαν τα ίδια πράγματα που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Η βασική έρευνα δεν μπορεί να δώσει άμεσα αποτελέσματα παρά μόνο μεσοπρόθεσμα, δεν μπορεί να αποδώσει άμεσα. Η βασική έρευνα δεν μπορεί παρά να χρηματοδοτηθεί από τον δημόσιο τομέα. Δεν έχει σημασία να συγκρίνουμε την χρηματοδότηση της βασικής έρευνας με τους βιομηχάνους που αναζητούν άμεσα το κέρδος. Θα πρέπει λοιπόν είτε είναι περιφερειακά τα χρήματα είτε εθνικά είτε κοινοτικά να στρέφονται στη βασική έρευνα. Δεν μπορούμε να ζητάμε λοιπόν αποτελέσματα από την βασική έρευνα. Είναι προφανές αυτό. Πρέπει να βρεθεί κάποιος απλός τρόπος που να επιτρέπει τους ερευνητές, στους ερευνητές να ερευνούν. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε εδώ κάποιες δυσκολίες ε, οι οποίες έχουν ήδη υπογραμμιστεί και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί η Ευρώπη σήμερα έχει αρχίσει να την ξεπερνά θα έλεγα η έρευνα από άλλες χώρες. Θα βρεθούμε πίσω από την Κίνα και από άλλες αναδυόμενες οικονομίες. Πρέπει να δούμε το πρόβλημα λοιπόν σοβαρά και πρέπει να δημιουργήσουμε κανονισμούς που να μην είναι εμπόδια αλλά πλαίσια. Πράγματι δύο γαλλικές λέξεις, ε, ρεγκλεμό, κανονισμός και καρκό, καύκος λοιπόν. Πράγματι η προσπάθεια αυτή την οποία ξεκινήσαμε έχει ενδιαφέρον και δεν αφορά αποκλειστικά στην έρευνα και εδώ δέχομαι ότι η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική αλλά εφαρμόζεται και στα ταμεία συνοχή, στα διαφορετικά ταμεία και στην γεωργία ότι επηρεάζει και τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες από έναν μικρό δήμο μέχρι τους γεωργούς, τις αγροτοβιομηχανικές μονάδες. Μιλάμε δηλαδή για ένα φαινόμενο σφαιρικό και όχι κάτι το οποίο είναι, δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει αποκλειστικά στον τομέα της έρευνας. Στην περίπτωση πάντως του τομέα της έρευνας, ακριβώς τα πλαίσια κάποιων προσπαθειών απλούστευσης ε, συνειδητοποιήσαμε ότι έχουμε κάποια θέματα, είδαμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο έχει, έχει παρέμβει ε, για να μπορέσει να βοηθήσει, να δούμε ακριβώς ε, τι γίνεται με κάποιες συνεργασίες και μορφές χρηματοδότησης και με πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν το είναι το θέμα να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ε, blame and shame, να, δεν αναζητούμε να, να ονοματίσουμε μόνο κάποιους οι οποίοι μετέχουν σε διαδικασίες που δεν εξελίχθηκαν καλά αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι διαφεύγουν του ελέγχου. Άκουσα κάποιους ομιλητές να λέγουν ότι ε, εμείς καλύπτουμε ένα μεγάλο ποσοστό των δαπανών μας χωρίς κανένα έλεγχο ε, λογιστικό και μάλιστα και σε τομείς οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί όπως το κοινωνικό ταμείο. Φυσικά απαιτείται απλούστευση, αλλά όχι μόνο για ένα συγκεκριμένο τομέα, αλλά γενικότερα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και τα δρακόντια μέτρα τα οποία ισχύουν μερικές φορές δεν διευκολύνουν τα πράγματα παρά μόνο κατόνομα. Συνεπώς λοιπόν Ακούμε με ανησυχία και έκπληξη αυτά τα οποία είπε κάποιος από τους ε, προλαλήσαντες ε, για το Ινστιτούτο Max Planck σαν παράδειγμα ότι δεν μπορείτε να πάρετε δάνεια, δεν μπορείτε να δανειστείτε χρήματα. και τέτοιου είδους ε, μορφές ενίσχυσης. Νομίζω ότι είναι ένα χρήσιμο στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη και δεν είναι το μόνο. Είμαστε όμως ανίκανοι να βρούμε μια λύση, είμαστε ανίκανοι να καλύψουμε το θέμα αυτό. 40 Λοιπόν, ε, θα πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος να είναι σχετικά σύντομος και ο οποίος να είναι αναγνώσιμος από όλους. Και το λέω αυτό και προς τον κύριο Τσάιλτς. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, όχι μόνο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτούς που παίρνουν τα χρήματα, αλλά μία εμπιστοσύνη ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους Το θέμα δεν είναι μόνο ότι χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα, το θέμα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης. Πιστεύω λοιπόν ότι η δυνατότητα η οποία υπάρχει ε, να συνεργαστούμε και με το ελεγκτικό συνέδριο έτσι ώστε σε όλες αυτές τις φάσεις ελέγχου και εξάντε και εξπόστ να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια θα έλεγα ρύθμιση εμπιστοσύνης έτσι ώστε να υπάρχει μία μορφή ελέγχου κάθε φορά στην κατάλληλη κλίμακα, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε τοπικό επίπεδο, αλλά που να είναι κάτι το σύστημα αυτό έμπιστο και πλήρες και σχετικά τώρα με την χρηματοδότηση ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία εγώ κατάλαβα αυτά τα οποία είπαν οι ομιλητές είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε έτσι ώστε αυτή η διατύπωση ε, των προϋπολογισμών μέσω των αποτελεσμάτων να προσαρμόζονται στις δραστηριότητες αυτών που ωφελούνται όχι μόνο στην έρευνα υπάρχουν προβλήματα, αλλά να δούμε και ποιοι άλλοι τομεί είναι αυτοί όπου η λογική αυτή της, ε, του προϋπολογισμού μέσω των αποτελεσμάτων είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες δυσκολίες. Νομίζω ότι είναι σαφές πάντως ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιάζουμε κάποια αποτελέσματα στους πολίτες οι οποίοι χρηματοδοτούν κάποιες δραστηριότητες, πληρώνουν κάποιες δραστηριότητες και πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται με τα χρήματά τους. Νομίζω εμείς ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτά έστω και με καθυστέρηση, έστω και σε διαφορετικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο όμως να το κάνουμε για να μην περιορίσουμε την δημιουργικότητα, την ελευθερία και την πολλαπλότητα της βασικής έρευνας. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει γιατί αλλιώς είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τα ωφέλη που μπορεί να έχει από αυτή την προσπάθεια. Θα ζητήσουμε τώρα από τους υπόλοιπους συναδέλφους, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση, δεν βλέπω κάποιον που θα ήθελα να πάρει το λόγο. Α. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Ε, δεν ε, έχω βέβαια προχειρές λύσεις, αλλά κάποιες ιδέες τουλάχιστον. Όσον αφορά τα λογιστικά συστήματα, ίσως είναι ε, στο λάθος τρόπος να αναφερόμαστε σε αυτά τα συστήματα ως λογιστικά συστήματα. Ίσως καλύτερο και πιο εφικτό θα ήταν να προσδιορίσουμε τις απαιτήσεις ε, σε ποιοτικές, ε, ε, σε, με ποιοτικά στοιχεία, να μην λέμε ότι πρέπει να ακολουθήσετε πούμε, το γερμανικό σύστημα ή κάποιο άλλο σύστημα, πώς ακριβώς θα θέλαμε να μεταχειριστούμε, για παράδειγμα, την, τις επενδύσεις, τότε μπορεί ο καθένας να δει το δικό του λογιστικό σύστημα και να δει πώς μπορεί να συμμορφωθεί με αυτό που προτείνεται. Αντί να λέμε ότι από 15 λογιστικά συστήματα πρέπει να διαλέξουμε ένα και μοναδικό. Να λοιπόν μια ιδέα γι' αυτό. Όσον αφορά την χρήση των δανείων. Κυρία Πρόεδρε, Ξέρετε, τον Υπουργό Οικονομικών μας είναι πάρα πολύ αυστηρός ε, με τον έλεγχο του δημοσίου χρέους ε, και δεν θα επιτρέψει σίγουρα τη χρήση των δανείων ε, στο νομικό πλαίσιο. Αυτή είναι η απάντηση η οποία ενδεχομένως να μην σας ικανοποιεί, αλλά αυτό που είναι μάλλον σημαντικό για ερευνητικούς οργανισμούς, ειδικότερα οργανισμούς που ειδικεύονται στη βασική έρευνα είναι η ιδέα που ανέφερα. Υπάρχει μια επένδυση, γίνεται μια επένδυση στην έρευνα και η απόδοση αυτής της ε, επένδυσης δεν εμφανιστεί στη σου, στο δικό σου οργανισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή συνεχές εισόδημα για σένα που να είναι η απόδοση της επένδυσης. Δεν υπάρχει λοιπόν μοντέλο επιχειρηματικό ε, στο οποίο να μπορεί να βασιστεί, Γι' αυτό ακριβώς το δάνειο δεν είναι ο τρόπο να χρηματοδοτήσει κανεί την έρευνα, επουδενή, ειδικότερα αν είναι βασική έρευνα, ε, αν υπάρχει, είναι πολύ κοντά στην εφαρμογή, αν έχει πολύ επαφή με τον κλάδο των χρηστών, τότε ίσω να είναι διαφορετικά τα πράγματα. αλλά τουλάχιστον όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα, δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και Μία ερώτηση όσον αφορά τα, τα καταποκοπήν ποσά. Ε, εμείς μπορούμε να τα δεχθούμε, είδαμε το 50 προς 25%. Εμείς θα προτιμούσαμε να είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Από τη μία υπάρχει η μέθοδος απλοποίησης και από την άλλη πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους ε, επαφή με την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, αλλά στη... τελικά αυτό θα σημαίνει ότι κάποιοι δικαιούχοι που δεν έχουν αυτό το καταποκοπήν ποσό ε, των γενικών δαπανών, υπάρχει περίπτωση να χρηματοδοτούνται υπερβολικά. Βλέπω το πρόβλημα, αλλά δεν έχω λύση. Και ολοκληρώνοντας ε, με την τελευταία μου παρατήρηση, δεν προτείνω και πάλι λύση, αλλά ο, Μαν, Μανουέλ Καντ είπε κάποτε πόσο, όσο περισσότερους νόμους ε, κάνει κανείς, τόσο περισσότερα είναι τα ε, συμφέροντα. Ε, αυτό είναι κάπως που, κάτι που το έχουμε χάσει, δηλαδή αν μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε ε, τα κονδύλια με κάποια απόσταση, τότε δεν θα χρειαζόμασταν όλους αυτούς τους λεπτομερείς κανονισμούς. Ευχαριστώ. Μάλιστα στο 1 τέταρτο που μας ε, απομένει μπορούμε να ζητήσουμε λοιπόν από τους προσκεκλημένους μας ε, βάσει των ε, ερωτήσεων που έγιναν να μας πούν ποια είναι τα συμπεράσματα που εξάγουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις κυρίας Γκρέσλε, του κυρίου Τεντανό, του κυρίου της κυρίας Αγιάλα Σέντερ και τις ε, δικές μου ερωτήσεις, αλλά όσον αφορά την παρατήρηση που, που αναφέρατε μόλι, την παρατήρηση που κάνατε μόλις τώρα αναφερόμενο στα δάνεια και στην έρευνα, εγώ ε, όταν ήμουν εισηγητής για το ΕΦΣΥ ήταν σαφές ε, ότι η ερευνητική, τα ερευνητικά ε, ιδρύματα, ειδικότερα βασικής έρευνας, δεν είχαν πρόσβαση στο ΕΦΣΥ αν ήταν δάνειο και δεν υπήρχε δυνατότητα διάθεσης των ποσών. Οπότε, ξαναρχίζουμε, σας δίνω το λόγο με, τον, με τη σειρά που λάβατε το λόγο και κατά τις παρουσιάσεις σας. Ο κύριος Βάλπρεκ πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω. Ε, όσον αφορά ε, την ε, προπαρασκευαστική δράση έχουμε κάνει μια αξιολόγηση όσον αφορά την εκτελεστότητα. Λυπάμαι αν είχατε διαφορετικές ε, ε, απόψεις που ακούστηκαν από διάφορες γενικές διευθύνσεις. Εμείς στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών θέλουμε να έχετε μια ενιαία απάντηση και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Έχετε περιθώρια βέβαια. Ναι, εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Πρέπει όμως να έχετε και τα απαραίτητα μέσα, λέει ο πρόεδρος, ε, γιατί ε, όταν ε, λέμε κάτι σε έναν επίτροπο, πρέπει να ξέρουμε και τι ακριβώς, περί τίνος ακριβώς ομιλούμε. Ναι, Κοιτάξτε, ως προς τους διεθνείς εταίρους μας, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον ΟΗΕ, Πρέπει να σας πω ότι όντως ε, υπάρχουν πολλαπλοί έλεγχοι, προσπαθούμε να τους απλοποιήσουμε, προσπαθούμε με το ελεγκτικό συνέδριο από κοινού να δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να βασιστούμε στους ελέγχους που έχουν γίνει από τους εταίρους μας ε, όταν έχουν γίνει ε, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά ε, πρότυπα. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής, η κυρία, η ελέγκτρια, η κυρία Μπαρσονέ του ΟΗΕ έχει ένα σύστημα αξιολόγησης εξάντε που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε κατά πόσο οι κανόνες των εταίρων μας είναι ε, συμβατές με τους δικούς μας. Ε, υπάρχει πάντως ένα κόστος, υπάρχει πρόοδος, ε, δεν σημαίνει ότι όλα είναι άχρηστα, αλλά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πάρα πολύ απλούστευση ακόμη να κάνουμε στον τομέα αυτό. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, ε, θα θέλαμε να ε, επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα όταν είναι δυνατό αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι η βασική έρευνα μερικές φορές δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο και σε αυτή την περίπτωση βεβαίως θα ε, συνεχίσουμε να δίνουμε επιδοτήσεις. Θέλουμε να έχουμε μια εργαλειοθήκη πλήρη που να μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση χωρίς να προβαίνουμε σε διακρίσεις. Αυτό το θέμα που έθεσε η κυρία Γιάλα Σέντερ είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να δίνουμε κατά αποκοπήν ποσά πολύ υψηλά σε έναν τομέα και καθόλου σε, ε, ε, και, σε άλλους τομείς καθόλου. Και πρέπει να φερνάμε λιγάκι και τους ελέγχους εξάντε. Φυσικά. Το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν τώρα. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ανεξάρτητο και γι' αυτό θα πρέπει ακριβώς να έχετε το δικαίωμα να πιέσετε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να τα αναγκάσετε να ομογενοποιήσουν τους λογιστικούς τους κανόνες και να πιέσετε και το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, γιατί το ποσοστό λάθους σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ μικρό, είναι εντελώς τυπικό ας πούμε στην ΚΑΠ, αρκεί να ξεχάσει κανείς ένα μικρό θάμνο κάπου για να θεωρηθεί ότι υπάρχει λάθος. Είναι πραγματικά παράλογο λίγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. με λίγο να βλέπω ότι εφαρμόζονται διαφορετικά λογιστικά συστήματα. Τα διεθνή λογιστικά συστήματα έχουν καθολικό χαρακτήρα και θα έπρεπε να εφαρμόζονται παντού. Ένα παράδειγμα να σας δώσω για να διαπιστώσει κανείς τη συνεισφορά της των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τρόπος που χρησιμοποιείται ποικίλει από χώρα σε χώρα. Ε, Um, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να εναρμονίσει τις διαδικασίες όχι μόνο μέσω των λογιστικών συστημάτων, όχι μόνο μέσω των, της απλούστευσης, αλλά κυρίως μέσω της εναρμόνισης. Έτσι θα πετύχουμε την απλούστευση. Εμείς ε, θα προσβλέπουμε να είμαστε σε θέση έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε τα εθνικά πιστοποιητικά ελέγχου στις προσπάθειές μας. Ναι, μεν είμαστε υπέρ α, του, της μοναδικής διαδικασίας ελέγχου, αλλά πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα εθνικά πιστοποιητικά ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα επίπεδα. Συνεπώς λοιπόν Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνεισφέρει τα μάλα δημιουργώντας ακριβώς τις ορθές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα πρέπει να είναι υποσυνεχή παρακολούθηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαζάρου. Θα συνεχίσουμε τώρα με την κυρία Ματανέ. Θα απαντήσω για τα χρηματοδοτικά μέσα και μετά ο συνάδελφος θα μιλήσει για τα καταποκοπήν. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι ότι μετά uh, Σχετικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν ε, ε, για το ΕΦΣΙ βλέπουμε και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δούμε τι δυνατότητες έχουν τα RTOs να δούμε ακριβώ τι γίνεται με το σχέδιο Juncker. And what we uh, see is that it can be a very smart complement Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πραγματικά κάτι το πάρα πολύ θετικό για συγκεκριμένα βέβαια, για συγκεκριμένους κλάδους, ακόμα και για την εφαρμοσμένη έρευνα. Ένα τρίτο είναι από τη βασική έρευνα, ένα τρίτο προέρχεται από την ανταγωνιστικότητα και ένα τρίτο από την ίδια τη βιομηχανία Φρανχόφα. Συνεπώς λοιπόν ακόμα και οι ιδιωτικές συμβάσεις για την εφαρμοσμένη ε, έρευνα ε, χρειάζονται κάποιες ε, επιδοτήσεις. Δεν έχουν απεριόριστες ικανότητες δανειοδότησης. Βλέπουμε λοιπόν τα εργαστήρια μας να χτίζουν κτίρια τα οποία υποστηρίζονται από τα διαφορετικά ταμεία και από δάνεια. Τα δάνεια αυτά απαιτούν όμως εγγυήσεις χρήσης και αυτή την εγγύηση μπορεί να τη δώσουν οι ε, μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι, συνεπώς λοιπόν ε, οι εγγυήσει που δίδουν είναι ότι θα χρησιμοποιούν τα κτίρια αυτά τουλάχιστον για τα επόμενα δέκα χρόνια και θα δαπανούν τα τόσα χρήματα. Αλλά για τις μικρομεσαίες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τέτοιου είδους ε, συμβάσεις. Και γι' αυτό η τράπεζα χρησιμοποιεί το θέμα της and δέουσας επιμέλειας ή της συμμόρφωσης. Γενικά υπάρχουν μέσα τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει και νομίζω ότι χάρη στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα έχουμε αρχίσει να το εξετάζουμε το θέμα. Βλέπουμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα όμως προς το παρόν δεν ανήκει αυτό το μέσο στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου αλλά ενδιαφέρει κυρίως την εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά δεν θα υπάρχει παντού στον κόσμο. Γνωρίζετε, λέει ο κύριος Αχτουή, ο κύριος εγώ έχω ζήσει την ιστορία του μεγάλου δανείου, εθνικού δανείου, ήμουν βουλευτής τότε δεν είχαμε την δυνατότητα να διαιτητεύσουμε ανάμεσα στις δαπάνες επένδυσης και στις δαπάνες λειτουργίας. Θυσιάσαμε δηλαδή τις δαπάνες επένδυσης και εφόσον δεν είχαμε πλέον χρήματα ε, εκδώσαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δάνειο. Αυτό είναι καρπός της μετριότητας διαχείρισης των δημοσίων χρημάτων. Λοιπόν, κλείνω το θέμα αυτό και περνώ στον επόμενο μιλητή. Σούτνα. Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω στο θέμα των ποσών κατά και το γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, τόσο μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά τα συστήματα λογιστικής. Γιατί οι πρωτογραφές είναι λίγο πολύ γνωστές και όλοι λίγο πολύ είναι κοντά στις διεθνές πρωτογραφές. Αλλά Υπάρχουν συγκεκριμένες μεθοδολογίε για να ανταπεξέλθουμε στι προδιαγραφέ. Και εκεί λοιπόν δεν υπάρχει σωστό ή λάθο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επίτευξη των προδιαγραφών αυτών. Το θέμα για παράδειγμα είναι το άμεσο κόστος. Δεν ορίζεται καθολικά ο όρος αυτός προκειμένου όλοι να καταλαβαίνουν ακριβώς το ίδιο σε ό,τι αφορά τη χρήση του όρου άμεσο κόστος. αν το λάβουμε λοιπόν αυτό υπόψη, βρισκόμαστε στην εξή κατάσταση. Το άμεσο κόστος από τεχνικής άποψης αποτελεί κάτι διαφορετικό σε διάφορες μεθοδολογίες. Μια μικρή οργάνωση ή μια οργάνωση που έχει σαφής διαχωρισμό μεταξύ των μονάδων μπορεί να παράγει πολύ πιο πολύ άμεσο κόστος στο σύστημα λογιστικής σε σχέση με μια αενοποιημένη οργάνωση που μοιράζεται το προσωπικό. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα ποσά καταποκοπή, Γιατί το ποσό κατά αποκοπή πώς ορίζεται. Η βάση υποτίθεται ότι είναι η ίδια για κάθε οντότητα. Προκειμένου να επιβάλλεται το ίδιο ποσό κατά αποκοπή συμπληρωματικά. Ο συνάδελφος του Μαξ Μάξ Πλάνκ είπε το εξή ότι αν τεθεί υψηλό ποσό κατά αποκοπή, ενδεχομένως ε, κάποιοι να μην μπορούν να ωφεληθούν λόγω τεχνικών ε, α, λεπτομεριών. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και πιο ενοποιημένες οργανώσεις, ε, περίπλοκες οργανώσεις με περίπλοκη υποδομή. Και υπάρχει και ένα σύστημα υπολογισμού του κόστους που, για παράδειγμα, λογιστική, μάλλον, το οποίο ενδεχομένω να υπολογίζει πιο πολύ α, το έμεσο κόστος. Το αποτέλεσμα φυσικά για το project είναι το ίδιο, απλά από τεχνικής άποψης καταχωρίζεται με διαφορετικό τρόπο. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα άμεσου κόστους και ε, πόσο κατά αποκοπή, ουσιαστικά επιταχύνεται αυτή η ανισορροπία, γιατί καταρχάς ε, το έμεσο κόστος το 100% και μετά προστίθεται και ε, το ποσό κατά αποκοπή. Και έτσι ουσιαστικά προωθούνται αυτοί που έχουν πολύ έμεσο κόστος. Και όπως είπε ο κύριος Έιλερ, έχουμε σε γενικές γραμμές αυτή την τάση για την ε, ενιαία ε, προσέγγιση και όπως όλοι ξέρουμε ε, αυτό δεν ισχύει ούτε για ερευνητικά προγράμματα ούτε για πουθενά άλλο ως σύστημα δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Να είσαστε σύντομοι γιατί όπου να είναι θα πρέπει να σταματήσουν και οι διερμηνείς. Ο κύριος Τόμα Εύθερμαν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να απαντήσω καταρχάς το ερώτημα για τα δάνεια. Ξέρουμε ότι σε επτά συστήματα τα πανεπιστήμια μπορούν να πάρουν δάνεια και σε επτά ε, συστήματα δεν μπορούν να το κάνουν παρά μόνο υπό αυτούς όρους. Επίσης, πιστεύουμε ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό πολλών συστημάτων δεν θα καθιστούσε πιθανή μια ενδεχόμενη αλλαγή αυτού γιατί πολλά συστήματα είναι υπό αυστηρό έλεγχο, προκειμένου ακριβώς να εντερηθεί αυτό το σύστημα. Και σε πολλές περιπτώσεις τα πανεπιστήμια εξακολουθούν να αποτελούν ιδρύματα δημοσίου δικαίου. Άρα δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει αυτό. Γι' αυτό αποκλεί μεγάλο αριθμό φορέων. Και τους αποτρέπει από τη χρήση τέτοια χρηματοδότηση. Ε, τέθηκε και ένα ερώτημα για την ε, πολυμορφία. Εμείς πιστεύουμε, και αυτό προέκυψε από όλες τις διαβουλεύσεις, είναι πολύ πολύμορφες οι ομάδες μας και ερευνητικέ ομάδες με μεγάλα πολλά ερευνητικά προγράμματα και ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλους που είναι εξειδικευμένοι σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ διαφορετικές οι ανάγκες τους και υπάρχει πιθανότητα να διαπιστώσουμε ότι τους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν του διαφορετικούς τύπους. Αυτό το ακούμε και από τις διαβουλεύσεις. όσοι δεν έχουν επαρκείς ικανότητες διαχείρισης και περνούν κυρίως από το εθνικό σύστημα και αυτοί κατά πάσα πιθανότητα θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν πιο πολύ τα ποσά κατά αποκοπή. Lump sums ή flat rates. Και είναι ενδιαφέρον γιατί διαπιστώνουμε ότι αυτοί που προτιμούν τα flat rates συχνά είναι από χώρε που δεν γνωρίζουν το πραγματικό κόστος των δραστηριοτήτων τους. Τρίτο σημαντικό σημείο. Όντως, η εικασία ότι ένα σύστημα πραγματικού κόστους θα ήταν πιο ακριβό από ένα σύστημα έμεσου κόστου, δεν στέκει. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από το project το οποίο υποβάλλει κανείς. Αν υπάρχει ένα project με υψηλό άμεσο για παράδειγμα υψηλό κόστο προσωπικού και χαμηλό κόστο υποδομών, το flat rate θα έδινε υπερβολική χρηματοδότηση ενδεχομένω. Αν υπάρχει ένα σύστημα με, χαμηλό, με χαμηλά έξοδα προσωπικού και ε, έμεσο κόστο ε, υποδομών που δεν μπορεί να εντοπιστεί, το ποσοστό αυτό αντιστρέφεται. Άρα, ω εκ τούτου, Νομίζω ότι και για τους χρηματοδότες καλό θα ήταν να επιτραπεί σε όσους έχουν σύστημα ελέγχου να το χρησιμοποιούν. Για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο υπήρχε μια θεωρητική δυνατότητα η οποία δεν λειτουργήσε, αλλά υπήρχε και προβλεπόταν θεωρητικά να ληφθούν υπόψη συστήματα πιστοποιημένα. Και εδώ στη συζήτηση αυτή είναι σημαντικό το εξή στοιχείο. Το θέμα δεν είναι αν θα υπάρξουν ε, διαφορετικά συστήματα πέραν του εθνικού. Θα υπάρξουν. Το θέμα είναι κατά πόσο να ακολουθούν τα ίδια πρότυπα. Και το θέμα λοιπόν δεν είναι να πιστοποιηθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά το κατά πόσο θα τηρούν τα διεθνή πρότυπα. Και κοιτώ για παράδειγμα τα πανεπιστήμια. Που στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έχουν αναπτύξει συστήματα με τους εθνικούς ερευνητές για το πώς ε, θα καταγράφονται κάποια, κάποιες δαπάνες. Και πάντα υπήρχε το ερώτημα του κατά πόσον αυτό θα ήταν αποδεκτό. Γιατί ενδεχομένω. να εντάσσονταν και άλλες δαπάνες στο σύστημα αυτό, αν υπήρξε αν υπήρχε μια κατανομή, θα μιλούσαμε ενδεχομένω για 0,01 λεπτά Άρα θα υπάρχουν από εθνική πλευρά σίγουρα εθνικά, μάλλον ε, διαφορετικά συστήματα, αλλά είναι σημαντικό να γίνουν αποδεκτά. Όταν μας λέτε ότι κάποιοι δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν το κόστος αυτού το οποίο κάνουν, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τα μέσα να το ενθαρρύνουμε αυτό έτσι ώστε να αποκτήσουν την δυνατότητα να γνωρίζουν τι κάνουν. Πώς θα κάνουμε κάτι καλύτερο άμα δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις επιδοτήσεις σαν μόχλο έτσι ώστε να καταλήξουμε σε σωστές πρακτικές. Για τις μικρομεσαίες να πω ότι εγώ έχω δουλέψει 17 χρόνια στα, στα νοσοκομεία στο Παρίσι, 10 χρόνια στο Ινστιτούτο Παστέρ 7 χρόνια στο Νοβάρτης και τώρα σε αυτήν την μικρή αν θέλετε εταιρεία που λέγεται Φυραλής και κάθε φορά τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε σε σχέση με το έμεσο κόστος και τα λοιπά και την απόσβεση τίθενται με διαφορετικό τρόπο. Ε, για τις μικρομεσαίες τώρα θα ήθελα να πω οι λογιστικοί έλεγχοι δεν μας δημιουργούν πολλά προβλήματα και μιας και οι μικρομεσαίες παίρνουν, υφίστανται μάλλον πολλούς ελέγχους και σε εθνικό επίπεδο γιατί έχουν τύχει εθνικών μορφών στήριξης, πιστώσεων, ε, επιστρέψιμων σε περίπτωση επιτυχίας κτλ. Δεν δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα. Ακόμα και το FRS, ε, αν μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε παντού, αυτό θα ήταν κάτι το πάρα πολύ θετικό Νομίζω λοιπόν ότι οι πιστώσεις είναι χρήσιμες για τις μικρομεσές και για, όλες, και για όλα τα προγράμματα τα οποία συντονίζονται από τις ίδιες τις μικρομεσές. Νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την, την ποικιλότητα των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης στην Ευρώπη και θα πρέπει να ποικίλουμε ακόμα περισσότερο και να είμαστε πιο εφάνταστοι σε επίπεδο μικρομεσαίων. Έχουμε μικρό χαμηλό επιτυχία σε σχέση με τα παραδοσιακά προγράμματα που λαμβάνουν επιδοτήσεις κάτω από πολύ ενδιαφέρουσες μορφές, αλλά για τα δάνεια υπάρχουν κάποια διμερεί διεθνικά ανάμεσα σε δύο χώρες έχουμε ποσοστά επιτυχίας 30%. 40% ε, μας δίνουν φτερά για να πάμε πιο γρήγορα. Κοιτάξτε και θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την ύπαρξη της προστιθέμενης αξίας, όχι μόνο την διανομή των χρημάτων. Ε, τι γίνεται λοιπόν που ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός παρεμβαίνει είτε, παρεμβαίνει είτε με επιδοτήσεις είτε με δάνεια και χωρίς αυτές τις ε, παρεμβάσεις τα πράγματα δεν θα προχωρούσαν. Παρακαλώ να είστε σύντομος, έχουμε τρία λεπτά μόνο διερμηνίας ακόμα. Για όλα τα προγράμματα αυτά χρειαζόμαστε ε, την καινοτομία και δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρο αποτέλεσμα για όλα τα προγράμματα που διαχειρίζονται ε, οι μικρομεσαίες κοντά στην αγορά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται Όλες οι μορφές χρηματοδότησης και τα δάνεια είναι χρήσιμα για προγράμματα τα οποία είναι κοντά στις αγορές ή κοντά στην επαγγελματική πρακτική εφαρμογή τους. Καλώς λοιπόν τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρία σημεία. Καταρχά, η έρευνα που ανέφερα προηγουμένως όσον αφορά τον ορίζοντα 2020 έθεσε επίσης το ερώτημα του πώς ε, θα συγκριθούν ε, οι τωρινέ μα διαδικασίε με άλλα προγράμματα ενίσχυσης στον τομέα τον ερευνητικό. Και η μεγάλη πλειοψηφία όσων απάντησαν ε, των συμμετεχόντων μας είπαν ότι δεν έβρισκαν άλλα συστήματα ε, που να είναι απλούστερα, ευκολότερα ε, να τα διαχειριστεί κανείς. Αυτή, αυτές είναι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων μας. Είναι ένας δείκτης διαφορετικός από αυτόν που είχαμε στο παρελθόν. Δεύτερο σημείο. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε όσον αφορά την εναρμόνιση του συστήματος ε, του λογιστικού ε, στα κράτη-μέλη. Εν τω μεταξύ όμως προσπαθούμε να κινηθούμε προς μία αναγνώριση του συστήματος του λογιστικού ε, των συμμετεχόντων μας αντί να υπάρχουν παράλληλα συστήματα μόνο και μόνο για να εξυπηρετούν τις ανάγκες μας. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αυτό που δεν πρέπει είναι να υπάρχουν δύο... Ε, λογιστικές. Μία λογιστική πραγματική και μία άλλη για να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες πρέπει, ε, το, ε, πρέπει το, το, η πηγή να είναι ίδια. Ναι, συμφωνώ απολύτως λέει ο κύριος Τσάιλ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και γι' αυτό θεωρώ και το βασικό δίδαγμα νομίζω είναι μια ευρύτερη βούληση να κινηθούμε προς την κατεύθυνση του να βλέπουμε καλύτερα την επιπρόσθετη αξία την ε, προστιθέμενη αξία της δουλειάς μας και όχι να βλέπουμε απλώς το γραφειοκρατικό μας σύστημα και να προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Νομίζω ότι σε συλλογικό επίπεδο πρέπει να στοχεύουμε σε συστήματα που μπορούν καλύτερα να καταδείξουν το την προστιθέμενη αξία και τον αντίκτυπο των όσων κάνουμε. Η διαδικασία λοιπόν που μας οδηγεί στη διαχείριση μιας τέτοιας προσπάθειας ε, ε, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μία ε, προσπάθεια δημιουργική που πρέπει να γίνει από όλους μας. Πρόεδρος, ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη και πρέπει να δεχθούμε όλοι μαζί ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Πρέπει να είμαστε τολμηροί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να προοδεύσουμε. Η κυρία Γκρέσλε θα συνοψίσει. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό το mid-term revision, η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, ε, θα μας ε, ε, βρει απολύτως θα μας αφήσει απολύτως, απολύτως ικανοποιημένους. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και πλέον ε, μπορούμε να βασιστούμε στην εξέλιξη των πρακτικών στις διάφορες γενικές διευθύνσεις. Κύριε Γκρέσλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, ε, που, μας, ε, που μοιραστήκατε μαζί μας τη θλίψη σας και τις απόψεις σας. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε και να μην ξεχνάτε ε, ότι θα θέλαμε πραγματικά να έχουμε τα έγγραφα όλων όσων μας είπατε. Ε, θα μας βοηθήσει και μας και τους εισηγητές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Επιτροπή των Προπολογισμών και τον Πρόεδρο Αρτουή. Ε, γεια σας και καλό βράδυ.